to avoid the criticism of Sir Robert, we would start only with the... Κύριε Ρόμπερτ, μόνο δέκα λεπτά καθυστέρηση έχουμε. Μικρή, προσπαθούμε να βελτιωθούμε πάντως. Και πρώτο θέμα για την απογευματινή συνεδρίασή μας είναι η σύσταση στο, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως για τις διαπραγματεύσεις για τη στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Γέγκλε να λάβει το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σκιώδη συγκητέ, και συνάδελφοι που είστε εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, βοηθή γραμματής που μας έχετε βοηθήσει σε όλη αυτή την ιστορία. Μέχρι στιγμής μπορώ να πω με πολύ καλή συνεργασία και με τους σκιώδεις ηγητές και το προσωπικό μας, αλλά και συναδέλφους από τον Καναδά, από την αντιπροσωπεία του Καναδά, στην οποία συμμετέχω ως αντιπρόεδρος, ε, εξεργάστηκα το θέμα αυτό. Πέραν των ευχαριστειών που ήθελα να εκφράσω, θέλω ρητά να απευθυνθώ και στη γραμματεία των ομάδων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να τους ευχαριστήσω για την υποστήριξη που μου έχουν προσφέρει για την ΕΕΔ. Θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετική η δουλειά, η συνεργασία που μου προσέφεραν. Μια συνεργασία η οποία πιστεύω θα μας επιτρέψει να έχουμε μια καλή ε, ένα καλό αποτέλεσμα της εργασίας μα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βιομηχανικό κράτος, ο Καναδάς, ο εκ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη, πολύ σημαντικό εταίρος και στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, αλλά και, και εδώ έχουμε τη μεγάλη σημασία αυτή τη συνεργασία, τα οικονομικά ζητήματα. Στρατηγικές λοιπόν και σημαντικές αλλά και πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, στις οποίες θέλουμε να δώσουμε μία νέα ε, μορφή, ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αρμόζει και στις ισχύουσες την επικαιρότητα συνθήκες, δηλαδή μια συμφωνία στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Η βασική ε, συμφωνία ανάγεται στο 1976. Δεν ξεκινάμε δηλαδή από μηδενική βάση. Έχουμε μια παλαιά συμφωνία, την οποία τώρα εξυγχρονίζουμε με βάση τις ισχύουσες συνθήκες και ανάγκες. Είμαι πεπισμένη ότι έχει ουσιώδη σημασία αυτή η συμφωνία για την πιο εντατική ε, συνεργασία, αλλά και για να έρθουν πιο κοντά και οι πολίτες των δύο πλευρών. Αυτή η συμφωνία μπορεί να τεθεί ενισχύ μόνο εφόσον εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εγκρίνουμε και ιδιαίτερος θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή μας αλλά και την Ολομέλεια να μεριμνήσει ώστε να γίνει και εγκαίρος αλλά και πλήρως η ενημέρωση ώστε να έχουμε μια πολύ καλή πλειοψηφία στην ψηφοφορία για την έγκριση όλες οι συμβατικές σχέσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Κρατών απαιτούν μια κοινή προσέγγιση. Αυτό ισχύει και για τα βιομηχανικά κράτη. Και βλέπω, πιστεύω ότι οι συμφωνίες ε, αυτές θα πρέπει να ε, καλύπτουν όλες τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Και πιστεύω ότι είναι προτιμότερη μια αυστηρή γραμμή, αυτό έχω επιλέξει, αυτό άκουσα να είναι και η προτιμόμενη προσέγγιση και από την πλευρά του Καναδά και από όσους ε, είχα την ευκαιρία να συλλομιλήσω. Και έτσι, εάν εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε να αποφασίσουμε ποια επιλογή θα, ποιο δρόμο θα επιλέξουμε για να διαφυλάξουμε και την αξιοπιστία μας για το μέλλον, με το κείμενο που έχουμε μπροστά μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγράφει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά και επιφυλάξεις με τη μορφή μιας συστάσεως προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις διαπραγματεύσεις. Και συνειδητά χρησιμοποίησα ευρείες αλλά και γενικές ε, διατυπώσεις, ώστε να έχουμε στο δυνατόν πιο ευρύ κατάλογο, θα έλεγα, ένα ευχολόγιο για να καλύψουν στο δυνατόν πιο πολλά θέματα και διατυπώνω και την, ε, το αίτημα για την ταχύτατη ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ένα σημείο το οποίο θα ήθελα συγκεκριμένα να αναφέρω είναι το σχετικό με την ε, συμφωνία για τη θεώρηση διαβατηρίων. Ξέρετε ότι ο Καναδάς απαιτεί για τους Ρουμάνους, Βουλγάρους και Τσέχους πολίτες ε, την θεώρηση διαβατηρίου. Ένα, μια κρεμότητα, ένα θέμα που συνεχίστε, που διορνίζεται, ένα θέμα το οποίο πρέπει να θίξουμε, σημαντικό θέμα, και υπάρχουν βέβαια άλλα δύο που θα πρέπει να συζητήσουμε, αλλά στη γενική ε, θεώρηση της υπόθεσης αυτής, της εταιρικής αυτής σχέσης, κύρια σημασίας για την ε, προώθηση και έγκριση με βρήτα την πλειοψηφία της συμφωνίας αυτής από το Κοινοβούλιο είναι η ρύθμιση του ζητήματος της θεώρησης διαβατηρίων. Με τους ε, σκιώδεις λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτατα και εγκαίρως οι διαβουλεύσεις, οι επαφές, η επικοινωνία ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό ταχύτατα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα ψηφοφοριών. Προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 18 Σεπτεμβρίου στις 10 Οκτωβρίου θα ξανασυζητήσουμε με τις τροπολογίες. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας προβλέπεται για τις 14 Νοεμβρίου και κατά πάσα πιθανότητα στο Στρασβούργο θα ε, δει το θέμα η Ολομέλεια τον Δεκέμβριο. Αυτά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και για άλλη μια φορά σκιώδη και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι μου ε, με βοήθησαν και τους παρακαλώ όποιος θέλει να συμβάλλει στην υπόθεση αυτή και να με στηρίξει αλλά και να μου υποδείξει σημεία που ενδεχομένως ε, σημειώνονται προβλήματα για να έχουμε στο δυνατόν πιο ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μοντάλ το παρακαλώ. Thank you very much. Um, I will try and be as brief. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι όσο σύντομος μπορώ. Όπως είπε και η συγκήτρια πρώτα απ' όλα, Δύο είναι συμφωνίες παράλληλες SPA και CETA και οι δύο σημαντικές και αξίζει να επικεντρωθούμε και να εστιάσουμε σε αυτές ε, για να ξαναδούμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Θα ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο. Τα εξής δύο μάλλον. Πρώτον, πολύ σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή συνάπτουμε συμφωνία μας Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Καναδά. Όλα τα κράτη-μέλη εντός της Ένωσης θα πρέπει να την χάνουν ε, ισότιμη μεταχείριση. Τι σημαίνει αυτό. Η αυτόματη άρση υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων για τους περισσότερους πολίτες των περισσότερων κρατών είναι γεγονός με εξαίρεση τη Ρουμανία, Βουλγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία. Για μας το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό να ε, το ξαναδούμε και απευθύνω μια έκκληση διακομματικά να υποστηριχθεί αυτό το αίτημά μας. Ε, αλλά και πέρα από κράτη-μέλη για να εκφραστεί πλήρης η αλληλεγγύη μας για το θέμα αυτό. Δεν θα ήταν δίκαιο να γίνει ε, συμφωνία στρατηγικής εταιρική σχέσης και να φεθούν αυτές οι τρεις χώρες ε, στην ισχύουσα κατάσταση. Εκτός εάν υπάρξει σαφής και μονοσήμαντη ένδειξη, και ποια ένδειξη, πολύ περισσότερο από ένδειξη θα πρέπει να είναι, ε, ότι θα ληφθούν εκείνες οι ενέργειες και θα γίνουν τα βήματα να ε, καταβληθεί αυτή η ανομαλία, διότι περί ανομαλίας πρόκειται. Δεύτερον, το συζήτησα και με εκπροσώπους της Καναδικής Αποστολής στις Βρυξέλλες και αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τη διατύπωση εκεί όπου αναφερόμαστε στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και τα συναφή. Εκείνοι τι λέγουν. Γιατί είναι σημαντικό να λέμε και τη δική τους άποψη, ακόμα και αν διαφωνούμε. Λένε λοιπόν ότι δεν ισχύει αυτό για την περίπτωση του Καναδά. Δεν είναι σωστή αυτή η διατύπωση. Γιατί ο Καναδάς είναι μια πλήρως ανεπτυγμένη δημοκρατία και δεν πρέπει να του φερόμαστε σαν να ήταν μια δημοκρατία ατελής ας πούμε. Η δική μας απάντηση ανέκαθεν έλεγε ότι Θα ήταν μάλλον διακριτική μεταχείριση αν χρησιμοποιούσαμε διαφορετική διατύπωση για διαφορετικές χώρες. Προφανώς θα πρέπει να γνωρίζουμε και δεχόμαστε ότι δεν έχουν όλες οι χώρες το ίδιο επίπεδο δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών. Αλλά από τη σκοπιά του Καναδά τουλάχιστον όταν το συζητήσαμε, ξεκαθάρισαν ότι η παρούσα διατύπωση δεν τους έβρισκε σύμφωνο και δεν ήταν διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση να τη δεχθούν. Διότι κατά την άποψή τους ε, αμφισβητεί τη δημοκρατικότητα της χώρας. Επισκιάζει κάπως. Από την άλλη, εμείς ως εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε την άποψη ότι είναι μάλλον δύσκολο να ε, αποστούμε από την ε, φυσική διατύπωση και ε, κανονική σε όλες τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης στρατηγικές. Είναι ένα τυπικό αυτό ε, και μια πάγια διατύπωση για όλες τις χώρες και δεν μπορούμε τώρα για τον Καναδά να αλλάξουμε ε, αυτή τη διατύπωση γιατί θα ε, σημαίνει αυτό διάκριση έναντι άλλων κρατών που δεν έχουν τόσο υψηλά κριτήρια δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Montalto. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μοντάλτο. Η κυρία Βέμπερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθεια που έχει καταβάλει και θα ήθελα να πω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά ήταν πολύ καλές και πρέπει να συνεχίσουν, να συνεχιστούν έτσι. Ο Καναδάς δεν είναι μόνο παραδοσιακός ε, εταίρος, αλλά μια δυνατή δημοκρατία. Έχουμε κοινά πολιτιστικά στοιχεία, τις ίδιες αρχές και αξίες. αξίες. Γι' αυτό είναι απόλυτα λογικό να συνεχιστούν αυτές οι σχέσεις, όπως ήδη έχουν διαμορφωθεί. Τώρα, ορισμένα σχόλια. Ένα θέμα που είναι πιο ευαίσθητο είναι πώς οι ε, Καναδοί ε, αντιμετωπίζουν ορισμένους ε, πολίτες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως Βούλγαροι και Ρουμάνοι καθώς και οι πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας που χρειάζονται θεώρηση για τον Καναδά. Θα υποβάλω μια τροπολογία και θα έρθω σε επαφή και με άλλους συναδέλφους για να υποβάλουμε ενδεχομένως μια κοινή τροπολογία. Όταν ε, ε, δούμε την στρατηγική συμφωνία από τη ε, πλευρά και τις εμπορικές συμφωνίες, την εμπορική συμφωνία, συμφωνία εμπορικών συναλλαγών από την άλλη, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε να έχουμε λίγο πιο δικονομική προσέγγιση. Εμείς ασχοληθήκαμε με τη στρατηγική συμφωνία εταιρικής σχέσης, η ίντα με το άλλο σκέλος με τις εμπορικές συναλλαγές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει ερεσιμότητα ε, στη Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή της δεύτερης. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εντελώς αυτόνομες αυτές οι συμφωνίες και ίσως να βρούμε και μία διατύπωση προς αυτή την κατεύθυνση. Θα υποβάλω και σχετική τροπολογία ως προς τη ρήτρα περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικά αυτή την ε, προσέγγιση που θέλουμε να ενταχθεί στη Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να δούμε και τις ε, αρχές μας, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να, και, να είμαστε και δίκαιοι ως προς τη διατύπωση που προβάλλουμε όταν μιλάμε για τέτοιες ε, ρήτρε. Δεν θέλουμε να στρώσουμε, να ανοίξουμε ένα ε, δρόμο συμφωνίας με τον Καναδά. Υπάρχουν ε, πολλά είδη συμφωνιών ανά τον κόσμο και δεν νομίζω ότι ο Καναδάς ε, ε, θέτει προβλήματα σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, εν πάση περιπτώσει, η τροπολογία μου θα έχει μια ειδική διατύπωση που θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική ως προς αυτό το θέμα. Η κυρία Σουίκα, η Σουίσα, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω όλους για αυτές τις κοινέ προσπάθειες που καταβάλλονται έτσι ώστε να υποβληθεί αυτή η πρόταση ψηφίσματος και να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Ως νέο μέλος... Και επειδή συμμετέχω στην αντιπροσωπεία ε, σχέσεων μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω αυτή την πρόταση. Ευτυχώς πολλοί βρήκαν τη θέση που τους αρμόζει στον Καναδά, βρήκαν θέσεις εργασίας χωρίς να χρειάζονται θεώρηση. Αλλά δεν δέχομαι το σημείο H το οποίο είναι λιγάκι αμφιλεγόμενο και βλέπω ότι τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται θεώρηση για να μεταβούν στον Καναδά. Υπάρχουν ε, οι συμφωνίες, συμφωνία εταιρικής ε, στρατηγικής σχέσης οι και οι ΣΟΕΣ, θα πρέπει όμως να υπάρχει συμμεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με τις θεωρήσεις. Δεν μπορούν να υπάρχουν ε, πρώτης και δεύτερης κατηγορίες, κατηγορίας πολίτες. Όταν μιλήσαμε για την ε, κατάσταση της Ένωσης στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα είπα ότι συμμεριζόμαστε όλοι κοινέ αρχές και θα πρέπει η μεταχείριση όλων των χωρών να είναι η ίδια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για χώρες βορρά και νότου, εντός και εκτός Σέγγεν και ούτω καθεξής πλούσιες ή φτωχές. Μιλάμε για κοινέ αξίες, δικαιοσύνη και δημοκρατία. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπονται αυτές οι διακρίσεις. Γνωρίζω βεβαίως ότι το επίπεδο δημοκρατίας δεν είναι ε, το ίδιο σε όλες τις χώρες. Αυτό αφορά και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μας, αλλά θα πρέπει να εναρμονίσουμε αυτά τα κριτήρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και θα υποστηρίξω τις, ε, την τροπολογία που θα αναφέρει ότι οι Βούλγαροι, ε, Ρουμάνοι και Τσέχοι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καθεστώς ε, θεωρήσεων. Ο Σε Ρόμπερτ. Πρόεδρε, δεν γνώριζα κάτι για το θέμα εκ των προτέρων. Μου έκανε εντύπωση αυτά που είπε ο συνάδελφος Μοντάλτο σε σχέση με, με το θέμα της γλώσσας. Συμφωνώ μαζί του. Εάν αμφισβητούμε τη δημοκρατία του Καναδά που είναι μία από τις καλύτερες του κόσμου, αυτό θα με εξέπλητε. Και αν δεν μπορούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε μια τέτοια συμφωνία, τότε δεν τα καταφέρνουμε καθόλου καλά. Νομίζω λοιπόν ότι αν είναι θέμα καθαρά διατύπωσης που δημιουργεί κάποια ανησυχία στους Καναδούς, τότε θα πρέπει να είμαστε αρκετά ευέλικτοι και να αλλάξουμε αυτή τη διατύπωση και να συμβαδίσουμε με τους ε, Καναδούς. Αυτό είναι το, το μόνο λογικό και δεν βλέπω που έγκυται το πρόβλημα. Πέτερλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ τάσομαι υπέρ των όσων προελέχθησαν. Ε, είμαι εισηγητής για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας και υπάρχουν θέματα που είναι παρόμοια με αυτά που μας απασχολούν εδώ, όπως τα προανέφερε η κυρία Βέμπερ. Θα ήθελα η, κυρία Βέμπερ να υποβάλει την τροπολογία της για να επιτύχει αυτό που αυτό που επιθυμούμε όλοι. Θα πρέπει να μην υπάρχουν διφορούμενα και παρερμηνίες από τους εταίρους μας. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, δείξουμε και εμείς την ίδια ευαισθησία με βάση τη δική τους ε, ευαισθητοποίηση ως προς το θέμα. Συμφωνώ λοιπόν ως προς το ότι εστιάσαμε την προσοχή μας πολύ σωστά στο όλο ζήτημα. Μιλάμε για τρίτες χώρες στην πρόταση ψηφίσματος. Γιατί η ορολογία, αυτός ο όρος δεν με καλύπτει. Εγώ θα μιλούσα για άλλες χώρες, λοιπές χώρες, όχι για τρίτες χώρες. Δεν τη βρίσκω, δεν βρίσκω ιδιαίτερα ευτυχή αυτό τον όρο, γιατί οι χώρες αυτές δεν θα συμφωνούσαν αν κατονομάζονται ως τρίτες χώρες και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κυρία Γέγκλε. Α, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Τάνοκ, ευχαριστώ πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Έχω και άλλη συνεδρίαση που έπρεπε να πάω. Δεν ήμουν στη συζήτηση παρόν. Η ομάδα μου θα κάνει τροπολογίε και μάλιστα σειρά τροπολογιών, συμφωνώ με τον κύριο Άτκιν για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Αυτό το μοντέλο ε, ενό μεγέθου που με αλαζονία έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι όλων των τρίτων χωρών όπω ονομάζει, ε, και συμπεριλαμβάνει και γνήσιες δημοκρατίες όπως είναι ο Καναδάς και η Ινδία. Και πραγματικά, αν μη τι άλλο, θεωρείται ως αλαζονική, όσο και απαράδεκτη στάση απέναντι σε χώρες όπως ο Καναδάς. Λες και ήμασταν εμείς οι διαιτητές για το τι στη δημοκρατία και ποιος έχει δικαίωμα και ποιον συνδέουμε με συμφωνία και έχουμε και δικαίωμα να ε, αναστέλουμε τη συμφωνία όταν φρονούμε ότι ε, δεν είναι δημοκρατικές. Δεν είναι δυνατόν να χάσουμε χώρες όπως είναι ο Καναδάς. Θα ήταν τραγωδία ε, όχι μόνο για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Και εγώ θέλω το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην έχουμε ε, αποκλεισμένες ε, χώρες από την κοινοπολιτεία. Αυτό το χρησιμοποιούν οι αντιευρωπαϊστέ όσοι θέλουν να φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο και σου λέει θα πάμε να ενωθούμε με τι Ηνωμένε Πολιτείε, τον Καναδά και άλλε χώρε τη κοινοπολιτεία. Η Βρετανική αντιπροσωπεία εδώ θεωρεί ε, πάρα πολύ ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε το ίδιο μοντέλο και την ίδια διαδίπωση προ όλου, γιατί τελικά ε, θα μείνουμε χωρί συμφωνία με συνέπειες ε, και ανεπιθύμητε και απρόβλεπτε. Ευχαριστώ κυρία Γέγκλε, παρακαλώ για να ολοκληρώσετε. Για να συνοψίσετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω ε, και να πω σε όλους που δεν ήταν παρόντες στην αρχή και δεν άκουσαν τα όσα είπα εγώ, να επαναλάβω και πάλι ξεκάθαρα ότι είμαι πρόθυμη να ακούσω όλες τις παρατηρήσεις σας, αλλά στο τέλος παρακαλώ θα πρέπει να έχουμε μία κοινή βάση για τη συμφωνία και δεν θα πρέπει να μας προσανατολίζει μόνο η συμφωνία με τον Καναδά. Σήμερα είναι η πρώτη και μόνο συζήτηση, θα διευρυνθεί η συζήτηση και σε άλλες χώρες με τις οποίες συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες και αυτές τις ευρύτερες συμφωνίες και τις γενικότερες. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Να δούμε μέχρι πού μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί, αλλά μετά κάποια στιγμή θα πρέπει να τεθεί και ένα τέρμα. Και θα παρακαλούσα ήδη από τώρα να μην ε, κάνουμε λόγο για αλαζονία όταν συζητούμε αυτά τα θέματα και λέμε ότι οικουμενικές μας αξίες, η η κοινή προσέγγιση που έχουμε εδώ, μπορεί να εμφανίζεται ή ενδέχεται να έχει τέτοια δράση σε κάποιες χώρες. Δεν είναι σκόπιμο όλα αυτά, ούτε αποτελεσματικά. Έχουμε και άλλες εμπορικές συμφωνίες. Βλέπε Νοτιοανατολική Ασία ή δεν ξέρω πού αλλού και βάσει αυτών εργαζόμαστε. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε και τις άλλες περιφέρειες και να έχουμε κάποια στοιχειώδη ε, ειλικρίνεια. Εγώ αυτό που δεν θέλω είναι να αποφασίσουμε κάτι το οποίο να ε, διακυβεύει και να αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία. Ε, δεν επιτρέπεται αυτό. Για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία μιλώνται ΣΟΕΣ. Γι' αυτό παρακάλεσα να συζητηθεί νωρίς αυτό το θέμα γιατί το περίμενα. Από το 2009 γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Καναδά και ε, συμφωνώ και με τους συναδέλφους που ε, έκαναν παρατηρήσεις για τη θεώρηση διαβατηρίων. Ο Καναδάς έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι πλήρης η άρση θεωρήσεων, αλλά έχει κάνει κινήσεις στην κατεύθυνσή μας. Και βέβαια ο Καναδάς έχει δικαιώματα και ανθρώπινα δικαιώματα και των μειονοτήτων και σε δημοκρατία ζει η χώρα, όπως και εμείς. Ε, ωραία. Και γιατί δεν μπορούμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία, δεν απαιτούμε τίποτα παραπάνω. Όταν λέει ο Καναδάς ότι μα και εμείς δημοκρατία είμαστε, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα και τα λοιπά. Ωραία, και πού είναι το πρόβλημα τότε για να υπογράψετε. Γιατί υπάρχουν προβλήματα με κάποιες μειονότητες, Πρόεδρε. Και τελειώνω λέγοντας, παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να τα διαβάσουμε όλα αυτά και να ασχοληθούμε με το θέμα πάρα πάρα πολύ εντατικά και με μεγάλη ακρίβεια, να δούμε τι τροπολογίες θα καταθέσουμε και σας παρακαλώ ειλικρινά να το ξαναδούμε, να το ξανασυζητήσουμε όσο θέλετε και να ε, βρούμε μια γραμμή, κύριε Πέτερλε, στραμμένη προς το μέλλον για κάθε συμφωνία, γιατί αλλιώς κάθε φορά θα δυσκολεύουμε τα πράγματα και θα είμαστε και ανηλικρινείς. Και εγώ δεν θέλω να είμαι. Θέλω να έχω μια σαφή βάση για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ρόιλ που είναι πρόεδρος Τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με την της Κορέα να μας ενημερώσει για την ε, επίσκεψή του στον Ιούλιο στη Βόρεια Κορέα. Στην Κορέα, σε αυτή τη χώρα της χαράς, σε βάση περιπτώσει. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με χαρά να σας ενημερώσω σύντομα για το ταξίδι μας 15 με 17 Ιουλίου Έχετε εκτενή παρουσίαση γραπτή στα χέρια σα, μπορείτε να τη διαβάσετε. Και αν θέλουν κάποιοι συνάδελφοι τη Επιτροπή Εξωτερικών επιπλέον ενημέρωση, είμαστε στη διάθεσή σα και εγώ φυσικά και όλοι οι συνάδελφοι που ήταν παρόντες. Επτά τον αριθμό μετέβησαν εκεί. Υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα και θέλω να το πω και εδώ. Θέλαμε να πάμε και στη Νότια και στη Βόρεια Κορέα, ω ήθιστε, αλλά λόγω τεχνικών ιδιαιτεροτήτων κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό μείναμε πάρα πολύ στη Βόρεια Κορέα και στη Νότια Κορέα είχαμε μόνο μισή μέρα και λίγο παραπάνω, τρία τέταρτα της μέρας. Αυτό μας ε, προκάλεσε προβλήματα γιατί οι Νότιο Κορεάτες ανησύχησαν που τους αφιερώσαμε τόσο λίγο χρόνο. Ε, πραγματικά με ευφύ συνομιλίες και τηλεφωνικές ε, λύθηκε. Η αποστολή αυτή γιατί έχει ενδιαφέρον για πρώτη φορά από το 2011 μετέβηκε πάλι την προσωπή υψηλού επίπεδου από την Ευρώπη στη Βόρεια Κορέα και μάλιστα σε ένα χρονικό διάστημα που η Βόρεια Κορέα ε, γνώρισε πολιτικές ε, δυσκολίες και θα γνώριζε αργότερα και, και τους ζήσαμε και αυτό ήταν πολύ τεταμένα τα πράγματα και η κατάσταση. Θα θυμάστε τις περίφημες απειλές από τη Βόρεια Κορέα ότι θα χτυπήσει με πυρηνικά λοιπά, Θα διακόψει τη συνεργασία, ότι θα κλείσει ε, το Κισόγκ, το ε, ε, βιομηχανικό αυτό συγκρότημα κτλ. Εμείς ουσιαστικά τι θέλαμε και το κάναμε και συνειδητά. Να έχουμε κάποιους διάβλους επικοινωνίας, να αρχίσουμε κάποιες επαφές, να αποκομίσουμε και εντυπώσεις, αλλά να δημιουργήσουμε και ένα πεδίο συνεννόησης. Στις συνομιλίες που είχαμε, πρέπει να πω ότι και στη Νότια Κορέα και στη Βόρεια έγιναν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, με τη Βουλή τους, με την ομάδα φιλίας, με τον ε, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, με τον Πρόεδρο της Βουλής και με εκπροσώπους επίσης μη κυβερνητικών οργανώσεων που διοργανώσαμε ήδη και ε, οργανισμούς του ΟΗΕ στην Pyongyang. Ενδιαφέροντα ήταν όλα αυτά, αλλά και οι επίσημες συνομιλίες. Είχαμε πάντα το ίδιο μοντέλο ε, επικοινωνίας, τίποτα καινούριο, τα πυρηνικά προγράμματα ε, η διακοπή τους θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για να ξαναγίνουν συνομιλίες και επίσης οικονομικές ε, συνομιλίες και η άση του μποϊκότ προϋποθέτουν να αλλάξει λίγο η εξωτερική τους πολιτική. Τι είπαν οι Βόρειο-Κορεάτες, προσπαθούσαν ανέκαθεν να τονίσουν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για αυτή τη δύσκολη κατάσταση και το έβλεπα λίγο διαφορετικά από εμάς ε, αυτό επαναλαμβανόταν κάποιες φορές και μέχρι που τους είπαμε ότι δεν μας βοηθάνε τώρα αυτά τα εθιμοτυπικά που μας λέτε, ούτε τον κόσμο στη Βόρεια Κορέα, ε, που δεν είναι και πάρα πολύ κατάσταση του. Και είδαμε πώς έχει και η στέγαση και τι κατάσταση επικρατεί, πώς ζουν οι καθημερινοί άνθρωποι σε αντίθεση με τα δημόσια κτίρια ε, που είναι πολύ εντυπωσιακά. Αλλά τα γνωρίζουμε σε τέτοια διαρθρωμένα συστήματα, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Στην αρχή του ταξιδιού είδαμε και στο Πεκίνο εκπροσώπους ε, της Κίνας με τον Βαντουβάη, ε, που είναι εκπρόσωπος της Κίνας στην εξαμερή διάσκεψη, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι και η κινέζικη πλευρά τα βλέπει κάπως διαφορετικά πλέον τα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν και αυτό ήταν ενδιαφέρον για τους συναδέλφους που πήγαιναν για πρώτη φορά. Είδαν ότι αλλάζει λίγο η στάση και της Κίνας. Έχει εκφράσει τη δυσφορία της για αυτά που κάνει η Βόρεια Κορέα. Και επίσης κάπου τόνισε ότι και η Κίνα έχει λιγότερη, μικρότερη δυνατότητα επιρροής ε, στη Βόρεια Κορέα από ό,τι σκεφτόμαστε εμείς ή η Δύση γενικότερα. Κάτι άλλο που είχε ενδιαφέρον στη Βόρεια Κορέα ήταν οι συναντήσεις που είχαμε με τους εκπροσώπους. Σας είπα ότι πάνω κάτω ήταν στάνταρ αυτά που μας έλεγαν, αλλά με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, οι συζητήσεις που έγιναν τυχαία και τους είδαμε στην αντιπροσωπεία του ΟΗΕ και είδαμε ποια έργα κάνουν και ποια επιτυχία και όχι μόνο αυτό, ότι τα διεθνή αυτά έργα των ΜΚΟ αφήνουν και αποτέλεσμα. Και όσοι εργάστηκαν εκεί μας είπαν ότι έχουν ένα πρόβλημα και μια ερώτηση. Και ήθελα να το πω και αυτό. Πρώτον, από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί έχει επέλθει μια κατάσταση που δυσκολεύονται ε, να κάνουν εμβάσματα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους πρέπει να πηγαίνουν ήδη στην Κίνα στην τράπεζα και αυτό τους δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή. Και αυτό είναι πραγματικά ενοχλητικό και λυπηρό γιατί δεν ήταν καθόλου ο στόχος των κυρώσεων. Και η δεύτερη πληροφορία που μάθαμε ήταν ότι πραγματικά αυτά τα έργα και τα προγράμματα έχουν ενδιαφέροντα αντίκτυπο. Στη Βόρεια Κορέα είδαμε και ήδη με τα μάτια μας ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκεί, έργο, και όπως γίνεται παντού δημιουργούν επαφές ε, αυτά τα προγράμματα, καταστρέφουν κάποια ε, εικόνα που έχει ο άλλος για τον εχθρό του και βοηθούν και τους ανθρώπους τελικά. Και ε, ρωτήσαμε μήπως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Όχι μόνο δηλαδή στη γεωργία και στα τρόφιμα, αλλά και σε άλλους τομείς. Στην υγεία, Φερρυπίνη, στην παιδεία, να σκεφτούμε μήπως υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα. Γιατί απλούστατα κάθε Ευρωπαίος που είναι παρόν εκεί στη χώρα και υλοποιεί ένα πρόγραμμα έρχεται σε επαφή με τους πολίτες ε, της Βόρειας Κορέας οι οποίοι μαθαίνουν ε, λίγο περισσότερο την πραγματικότητα ε, μαθαίνουν ότι αυτοί που τους μαθαίνουν να είναι εχθροί τους είναι κάπως διαφορετικά και θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή και σε τέτοια προγράμματα και έργα. Ας πούμε, θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή με τους Βόρειο-Κορεάτες εκτός της Ευρώπης, εκτός Βόρειας Κορέας. Αυτά βέβαια είναι μακράς πνοής. Η επιστημιστική κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και μάλιστα ορισμένοι προβλέπουν επιδείνωση ακόμα μεγαλύτερη Γι' αυτό νομίζω ότι για μας είναι σημαντικό και εδώ να συνεχίσουμε τη βοήθειά μας. Στη Νότια Κορέα σας είπα ήταν πολύ σύντομη η επίσκεψη. Συνοψίζω. Ε, να σας πω, είδαμε τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα λέω σύντομα γιατί έχετε και εσείς βαρύ πρόγραμμα. Είδαμε και τους συναδέλφους της Εθνοσυνέλευσης. Ήταν και τέλεια διοργάνωση αλλά και τεράστιος ο ενθουσιασμός. Παρόλο που πήγαμε Σάββατο πρωί και το βράδυ φύγαμε. Ήταν ε, παρόντες όλοι με μεγάλο ενθουσιασμό, με μεγάλο ενδιαφέρον για συνεργασία. Δεν υπήρχε πλέον καμία δυσφορία, καμία ανετική διάθεση που σας είπα ότι είχαν λίγο ενοχληθεί επειδή πήγαμε τόσο λίγο στην Νότια Κορέα και θέλησαν να μάθουν τι εμπειρίες αποκομίσαμε και εμείς από τη Βόρεια Κορέα και πού υπάρχει δυνατότητα επιπλέον βοήθειας ή ε, άλλος τρόπος βοήθειας. Ο υπουργό Εξωτερικών μας έκανε θετική εντύπωση, ειλικρινή, ανοιχτή. Δεν τον ενδιέφερε να κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα, ούτε να ε, αποδώσει ευθύνες αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να διερευνήσει τρόπους επικοινωνίας, διάβλους, έτσι, νήματα επικοινωνίας να το πω έτσι. Δεν πήγαμε στο Κεσόγκ, γυρνάω πάλι στη Βόρεια Κορέα, σε αυτό το βιομηχανικό σύμπλεγμα, γιατί μας είπαν ότι είναι στην αρμοδιότητα του στρατού και τέρμα, δεν ε, τίθεται ερώτημα. Για μας αυτό ήταν δυσάρεστο, αλλά τι να κάνουμε σε τέτοιες χώρες, το λαμβάνουμε υπόψη, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Από την άλλη, διαπιστώνουμε με μεγάλη χαρά και πάλι ότι κάπως έχουν κινηθεί τα πράγματα. Σήμερα το πρωί το συζήτησα με τον Νότιο Κορεάτη πρέσβη εδώ στις Βρυξέλλες. Αύριο ε, επαναλαμβάνει τη λειτουργία του συγκροτήματος και στο μέλλον θα διευρυνθεί και θα επεκταθεί. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο ανταλλαγές Βορείου-Νοτιού Κορέας, η Νότια Κορέα καταβάλει προσπάθειες να κατασταθούν εκεί και διεθνείς εταιρείες για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να μην ε, μπορεί κατά το ένας ε, από τους εταίρους να το κλείνει. Την άλλη εβδομάδα θα συναντηθούν οικογένειες από τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα. Μικρές συναντήσεις είναι αυτές, περιορισμένες, αλλά επαναλαμβάνονται παρόλα αυτά, ε, ξαναρχίζουν κάτι κινείται, εν πάση περιπτώσει. Η Βόρεια Κορέα είναι μια χώρα περιχαρακωμένη. Ε, ο κόσμος δεν περνάει καλά οι άνθρωποι. Πάντως υπάρχουν και νέοι που είναι περίεργοι, που ενδιαφέρονται να δουν και παρά έξω, ε, θέλουν να συνάψουν επαφές και να γνωρίσουν κόσμο και να έχουν και πιο μακροχρόνια επίπτωση όλα αυτά. Τέλος, τον Οκτώβριο θα έρθει να μας δει ο πρέσβης της Βόρειας Κορέας. Στο Στρασβούργο θα έρθουν Ιανουάριο μια αντιπροσωπεία της Βουλής της Νότιας Κορέας και αν σας ενδιαφέρει μπορούμε να διοργανώσουμε και νέα συνάντηση. Αξίζει τον κόπο πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά και είμαι πεπισμένος ότι και άλλοι συνάδελφοι έμαθαν πολλά. Ε, αποκομίσαμε πολύτιμες εμπειρίες. Εγώ γενικά βαριέμαι να ταξιδεύω, <laughs> αλλά χάρηκα που πήγα στην ε, αντιπροσωπεία αυτή και ήταν και οι επενδύσεις που έγιναν και οι εντυπώσεις που μας άφησε πολύ σπουδαίες. Σε Ρόμπερτ. Πολύ εντυπωσιακή αυτή η έκθεση. Για να κάποια ερωτηματικά βέβαια, για όποιον δεν είχε, όπως εγώ, την ευκαιρία να επισκεφθεί αυτήν την υπέροχη χώρα και ρωτώ εάν ε, είναι ικανοποιημένος ε, και αν μπόρεσε να δει όσα ζήτησε. Γιατί γενικά δεν δίνεται αυτή η εντύπωση ως προς ε, τη διαθεσιμότητα της Βόρειας Κορέας προς άνοιγμα του κόσμου. κόσμο. Επίσης υπήρξε μια επίσκεψη δημοσιογράφου Βρετανού στη Βόρεια Κορέα, ο οποίο με κρυφή κάμερα μπόρεσε να περάσει τα σύνορα και να καταγράψει, χωρί να αντιληφθεί κανεί. και αυτό βγήκε βέβαια μετά στα Βρετανικά μέσα, ε, μεγάλη φτώχεια, ακραία φτώχεια και πάρα πολύ δυσμενείς συνθήκες κράτησης στις φυλακές. Τρίτον, Δεδομένου ότι έχουν εκφραστεί πολύ συγκεκριμένε απειλέ, ότι έχουν στραμμένου πυράβλου προ τι ΗΠΑ κ.ο.κ. Είχατε την ευκαιρία να εκτιμήσετε τη στρατιωτική ετοιμότητα, τις δυνάμεις, ε, ενδεχόμενες προετοιμασίες ε, από την πλευρά των βορειοκορετών. Και τελευταία ερώτηση, μάλλον ρητορική. θα, θα λέγατε ότι η άγνοια μέσα στην οποία ζουν οι Βορειοκορεάτες για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο είναι ευλογία μάλλον ή κατάρα. Ο κύριος Ρόιλ. Δεν σας κρύβω, δεν σας αποκαλύπτω το κανένα ε, μυστικό. Ήταν φυσικά μια δύσκολη επίσκεψη, ήταν μια επίσκεψη που μας ε, προσγείωσε σε πολλά πράγματα, σε πολλά σημεία στην πραγματικότητα. Δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε όσα θέλαμε να επισκεφθούμε γιατί έπρεπε να λάβουμε άδειε. Και βέβαια είμαστε αναγκασμένοι να υποταχθούμε στην προοπτική και τις επιλογές της κυβέρνησης της Βόρειας Κορέας. Αυτό δεν σας το κρύβω. Ούτε είναι κάτι το αξιοπερίεργο. Αυτό όμω το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα για, τους, για τα όσα είπαν οι συνάδελφοι που έχουν επισκεφθεί πολλέ φορέ στη χώρα, γιατί και μόνο ήταν η πρώτη φορά. Διαπίστωσαν λοιπόν οι συνάδελφοι ότι είναι κάπω πιο ανοιχτή η χώρα. Υπήρχαν άνθρωποι με κινητά στα χέρια. Κινητά που, που μπορεί ε, έχουν συνδέσει μόνο μέσα στη Βόρεια Κορέα. Δεν έχει σημασία όμω. Υπήρχαν τα κινητά και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένω είχαν διαβιούν σε αποτρόπιες συνθήκες ε, ε, φτώχεια, σπίτια που δεν θα διανοούνταν κανένας Ευρωπαίος να, να μπει μέσα και να μείνει, αλλά υπάρχει μια διαφορά στην αξιολόγηση της κατάστασης από τους ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί πολλές φορές στη χώρα. Λίγο πιο ανοιχτό, λίγο πιο πολύ διάθεση για ε, διαπραγμάτευση, λίγο πιο πολλά αυτοκίνητα, τεράστιες οδοί με λίγα αυτοκίνητα, αλλά υπήρχαν κάποια περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν από ό,τι λένε, εργοστάσια, αυτοματοποιημένα. και, παραγωγή σε τέτοια ταχύτητα που ήταν εντυπωσιακή, αν και τελικά δεν υπάρχει αρκετό υλικό για να δουλέψουν τα εργοστάσια αυτά. Βεβαίως και έχουν πάρα πολύ κόσμο και δουλεύει ο κόσμος στα εργοστάσια, τις μικρά στρατιωτάκια που δουλεύουν στις αλυσίδες παραγωγής, αλλά και βεβαίως είναι στρατιωτικοποιημένα τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι να δούμε εάν από τη θέση που βρίσκονται μπορούν να δείξουν κάποια δίθεση να μετακινηθούν. Έτσι λοιπόν το πρώτο ερώτημα είναι αν μπορούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να κάνουν τη δουλειά τους και δεύτερον εάν κάθε πρωτοβουλία δική μας από την Ευρώπη, δηλαδή από τις ΗΠΑ μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα σημείο επαφής και κάθε σημείο επαφής αποτελεί μια ευκαιρία να μιλήσουν ή να συνομιλήσουν οι άνθρωποι στη χώρα αυτή, οι πολίτες δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να τους αποκλείουμε διαπαντός. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε. Βεβαίω. Και πρέπει να σας πω ότι έγινε μια απόπειρα να μας πούνε «Μα δώστε μας, παραδώστε μας τα κινητά και κτλ». Διστακτικά ίσως, αλλά εμείς είπαμε «Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρόκειται να τα πάρετε». Από την άλλη βέβαια ξέραμε ότι τα κινητά μας δεν θα δουλεύανε, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Προσπάθησαν όμως. Ε, και όταν εμείς αρνηθήκαμε, έκλεισε το θέμα. Βεβαίως στην ε, ρητορική που χρησιμοποιείται πάντοτε καταγγέλλονται τα υπετιότητα ε, των Αμερικανών και των, ε, και των Νοτιοκορεατών. Ε, υπήρξε κάποια φορά που χρειάστηκε να σταματήσω τον ομιλητή και να πω ένα λεπτό, όλα αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Σε εξηγήσω γιατί έχετε άδικο και γιατί η κατάσταση είναι αυτή και γιατί οι Νοτιοκορεάτε ζουν καλύτερα από ότι οι Βορειοκορεάτε και όλα αυτά. Όλα αυτά όμω μπορούν να αλλάξουν. Και έτσι Ε, και έτσι φτάσαμε πολύ γρήγορα στην κουβέντα του πώς μπορεί να ξανανοίξει το κεσόν. Και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια αξιοπιστία, κάποια μονιμότητα σε αυτό το άνοιγμα, γιατί βέβαια δεν θα έρθει κανεί να δουλέψει, ούτε θα ρίξει Θα, αρχίσει κανεί μια επένδυση ε, από πλευρά τη Νότια Κορέα, αν υπάρχει ο κίνδυνο να πα να ξανακλείσει το εργοστάσιο στο ΚΕΣΟΝ. Έτσι λοιπόν, είχαμε την εντύπωση, την αίσθηση ότι κάτι καταλάβανε. Αλλά μέχρι εκεί. Κύριο Πάσκου. Και εγώ μπορώ να πω από πλευρά μου και να βεβαιώσω ότι είναι πολύ πιο ανοιχτά, ανοιχτή η κοινωνία, το καθεστώς από το 99 που εγώ το επεσκέφθη. Δεν υπήρχαν τότε κινητά. Αυτό ήταν. Και ξέρετε το ανέκδοτο ήταν δύο Δύο κανάλια έχει τηλεόραση. Το πρώτο ε, έδειχνε μόνο ο Κίμιλ Σουν και στο δεύτερο υπήρχε κάποιο με το χέρι, με το δάχτυλο προταμένο που έλεγε πηγαίνει στο πρώτο κανάλι αμέσω. Τα πάντα ήταν ε, κενά καταστήματα κτλ. Ε, ο κύριος Μοντάλτο όμως. Σας ευχαριστώ. Και εγώ επισκέφθην την ε, Βόρειο Κορέα, δεν ξέρω αν συμπέσαμε εν αγνία μας, αλλά κατά πάσα πιθανότητα. Ε, περιπτώσει, αυτό που βλέπω είναι ότι οι ίδιοι Βόρειο Κορεάτες έχουν μια πολύ διαφορετική νοοτροπία από αυτήν που θα διαπιστώσει κανείς οποιαδήποτε άλλη χώρα με αυταρχικό καθεστώς. γιατί για δεκαετίες ανατρέφονται, τους γίνεται πλήση εγκεφάλου και έτσι πραγματικά πιστεύουν ότι ισχύουν αυτά που τους λένε. Ακόμη κι αν αυτά που τους λένε φαίνονται τόσο απίστευτα για μας. Αυτό νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο κόσμος σχέση με τη Βόρεια Κορέα. Ότι αντίθετα με άλλες χώρες αποκλεισμένες από τον κόσμο υπάρχει κάποια μορφή επαφής, επικοινωνίας, ανταλλαγής με τον υπόλοιπο κόσμο. Ενώ στην περίπτωση Βόρειας Κορέας είναι μάλλον απίθανο κάτι τέτοιο. και αν υπάρχει επαφή με τον έξω κόσμο ευκαιρία μόνο υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Και αυτό μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια ανεπαίσθητη χαλάρωση στο καθεστώς η Κίνα δεν ελέγχει όσο, όσο πιστεύαμε ότι ελέγχει τη Βόρεια Κορέα, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Η Βόρεια Κορέα είναι τόσο διαφορετικό κράτος, τόσο διαφορετική χώρα, που είναι σχεδόν αδιανόητο για μας το να συλλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει πώς ακριβώς σκέφτονται οι Βορειοκορεάτες. Όταν μιλάμε για στρατό ενός εκατομμυρίου ανδρών, εγώ θα σας πω ότι είναι μόνο κλάσμα της πραγματικότητας, γιατί κάθε Βόρειο Κορεάτης, άνδρας ή γυναίκα, ανήκει στο στρατό, είναι στρατιωτικός. Άρα, αν μιλάμε για τον μεγαλύτερο ή τον τέταρτο σε μέγεθο στρατό στον κόσμο, αυτό σημαίνει και πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο κάθε πολίτης με κάποιον τρόπο υπηρετεί στρατιωτική θητεία και ότι είναι προγραμματισμένος να πιστεύει σε μία Κορέα Αυτή είναι η ακράδαντη πεποίθηση και διακήρυξη Και αυτό είναι μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει κανείς να αντιμετωπίσει και μεγάλη πρόκληση. Λόγω ακριβώς της βαθιά ριζωμένης αυτής νοοτροπίας και αντίληψης ε, σε, του κάθε ενός και κάθε μίας Βορειοκορεάτη ή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόιλ θα πρέπει να αποχωρήσει. Ο κύριος Στάνοκ όμως ήθελε να λάβει το λόγο αν μπορέσετε να μείνετε ακόμα δύο-τρία λεπτά κύριε Ρόιλ. Ναι πρόεδρε. Θα ήθελα στον, ε, από το, τον Μαλτέζο συνάδελφο να ρωτήσω. Ξέρουμε ότι είναι ένα σταλινιστικό ολοκληρωτικό καθεστώς τρόμου ε, η Βόρεια Κορέα με ε, απόλυτη παραγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων. Φαίνεται ότι ο νέος ηγέτης της Βόρειας Κορέας ε, έδωσε εντολή να εκτελεστεί σύντροφός του πρόσφατα και πολλά άλλα τέτοια. Ε, πώς λοιπόν νομίζετε ότι όλα αυτά που μπορεί να σας προσφέρονται ως νέα εντύπωση να είναι απλώς χειραγώγηση από πλευράς της, ε, του, του καθεστώτος. Εγώ προσωπικώ αρνούμαι να επισκεφθώ χώρες σοσιαλιστικές γιατί δεν είμαι διατεθειμένος να τους προσφέρω την νομιμοποίηση ώστε να παραμείνουν στην εξουσία ε, με την επίσκεψη την οποία μπορούν να διαφημίσουν στη συνέχεια ως υποστήριξη από πλευράς μου όπως άλλωστε δεν πηγαίνω και στο Ιράν. Λοιπόν πώς θα κρίνετε όλα αυτά κύριο Ρόιλ. Πολύ καλή ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που πάντα μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολεί, αλλά για να σας ε, αναφέρω ακριβώς αυτό που είπατε κύριε συνάδελφο, ότι υπάρχουν ακόμη περισσότερα επιχειρήματα υπέρ του ότι καλά κάναμε και πήγαμε. Ακριβώς, γιατί μόλις ακούσαμε ότι έγινε αυτή η εκτέλεση, αποστήλαμε και επιστολή στην ε, πρεσβεία εδώ, αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας και είπα ότι έλαβα αυτή την ενημέρωση για την εκτέλεση και παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε αν έχει συμβεί και γιατί. Έτσι είχα το δικαίωμα, με την επίσκεψη που είχα κάνει, είχα το δικαίωμα να, να απευθύνω την, την ερώτηση και να μου απαντήσει ο πρεσβευτής της Βόρειας Κορέας. Αυτή είναι η εντύπωσή μου λοιπόν. Και θεωρώ ότι ήταν καλό το ότι πήγαμε, ήταν σωστό το ότι πήγαμε, βοήθησε, αλλά πάλι όπως είπα βοηθάει σε απειροελάχιστο βαθμό. Πάρα πάρα πολύ μικρή συμβολή. Για τους Βεωρικορεάτες σίγουρα δεν έχουμε βέβαια τόση αξία και σημασία. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ε, αν θέλετε μπορείτε να αποχωρήσετε. Εμείς προχωράμε στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης που είναι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ και θα ήθελα ο κύριος Τάνοκ που είναι και ο εισηγητής να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και όπως γνωρίζετε περισσότεροι, δεν ήταν ε, εύκολη έκθεση για το Σαχέλ, διότι η Δυτική Σαχάρα που ε, απασχολεί το εντέταρτον της έκθεσης μιλά για τις ζωηρές ε, απόψεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πόσο διφορούμενο το ζήτημα. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για τροπολογίες, επειδή υπάρχει παραπληροφόρηση και σύγχυση, ότι θα πρέπει να σας δώσω ορισμένες διασαφήσεις για την δημιουργία αυτής της έκθεσης. Εδώ και χρόνια έχω μία στεναρή στάση σε σχέση με τα δικαιώματα των Σαχαράουι στην περιοχή του Σαχέλ. Δεν ξέρω πώς θα είναι η τελική έκβαση του ζητήματος, αλλά ποτέ δεν θέλησα να περιλάβω τη Δυτική Σαχάρα στην έκθεση. Όταν δέχτηκα την έκθεση, θεώρησα ότι πρέπει να ασχοληθώ με την περιοχή του Σαχέλ. Κατέστη σαφές όμως ότι η Δυτική Σαχάρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης και η αρχική πρόταση των σοσιαλιστών ήταν να λάβουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Δυτική Σαχάρα. Φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό, λαμβάνοντας υπόψη και τη Δυτική Σαχάρα και την περιοχή του Σαχέλ, αλλά αυτό κατά της δικής μου ε, θέλησης. Δεν ήθελα να συμπεριληφθούν και τα δύο. Μετά από διαπραγματεύσεις ε, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει στον τίτλο να μιλάμε μόνο για την περιοχή του Σαχέλ και όχι την Δυτική Σαχάρα, αλλά η ΑΦΕΤ και η Ντρουά δέχτηκε την συμπερίληψη της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό το δέχτηκε και η διάσκεψη των Προέδρων. Ε, σε αντίθεση πολλές ε, κυβερνήσεις, εγώ υπέβαλα μία τελική πρόταση με βάση τη θέση της διάσκεψη των Προέδρων η Δυτική Σαχάρα είναι μια ξεχωριστή συζήτηση, αλλά αν λάβουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και την γεωπολιτική κατάσταση, θα πρέπει να γνωρίζουμε, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, θα πρέπει να υπάρχει μια ε, γενικότερη στρατηγική για την περιοχή του, του Σαχέλ. Σε αυτή την Επιτροπή λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια είναι ε, αδιαχώριστα ζητήματα. Υπάρχουν πολλοί καταβλισμοί στη Δυτική Σαχάρα και μία ε, τροπή προς την βία. Αν αφήσουμε τη Δυτική Σαχάρα κατά μέρος, θα ήθελα να λάβουμε υπόψη τις πέντε χώρες ε, της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαχέλ. Και ασχολούμαστε με τη μεγάλη καταστροφή στο Μαλί και στις χώρες της ε, Δυτικής Αφρικής, όπου πριν υπήρχε πολιτική σταθερότητα. Αν και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι η κρίση, την, την κρίση την έχουμε αντιπαρέλθει, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες και εσωτερικά ε, μετατοπιστέντες, ιδιαίτερα στο Μαλί. Και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, ζητήματα της περιοχής και όχι μόνο του Μαλή. Η συμφιλίωση δεν θα ισχύει αν δεν υπάρχει αντιστάθμιση. Το Μαλή θα πρέπει να είναι ένα πρότυπο για την δημιουργία ενός κράτους δικαίου. Δυστυχώς ε, τα εγκλήματα και ε, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας έχουν περάσει ε, Γι' αυτό ο Χισένε Χαμπρέ θα πρέπει να καταδικαστεί και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να λάβει θέση. Πέρα από το Μαλί και το γεγονός ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία, τόνισα την ανάγκη μια συνεκτικής στρατηγικής στη Σαχέλ, στην περιοχή του Σαχέλ για να προωθήσουμε την ασφάλεια και να ασχοληθούμε και με θρησκευτικά ζητήματα, να μην υπάρχει δουλεμπορία και εμπόριο ε, ναρκωτικών, ιδιαίτερα στους αυτοκινητοδρόμους της περιοχής του Σαχέλ και να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και την λογοδοσία του κράτους. Η έκθεση τονίζει την αποκέντρωση εξουσίας και το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Τέλος, ασχολούμαι με θέματα γυναικών, ιδιαίτερα τον ε, ακροτηριασμό των γυναικών και ιδιαίτερα την περίπτωση της καλαβιάς της ε, δούλεμπορίας στη Μαυριτονία. Κάτι το οποίο δεν δέχονται οι μαυριτανικές αρχές. Οι συμβιβασμοί που αφορούν τις πέντε χώρες του Σαχέλ έχουν ε, προωθηθεί αλλά σε πολλούς συμβιβασμούς ε, έχουμε εντάξει τροπολογίες από τη δεξιά μέχρι την αριστερά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοδομητική σας τάση και ως προς τη Δυτική Σαχάρα η κατάσταση ήταν πιο περίπλοκη. Έχουμε τροπολογίες συμβιβασμού για να, δεχτούν, να γίνουν αποδεκτές από όλο το πολιτικό φάσμα. Αρχικά είχαμε επιτυχίες αλλά δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες πολλοί συνάδελφοι ζήτησαν να αποσυρθούν τώρα από τους συμβιβασμούς. Με τους σκιώδεις είπαμε ότι θα πρέπει να δεχτούμε προφορικές τροπολογίες και στη συνέχεια να τις ε, καταψηφίσουμε. Αυτό σημαίνει όμως καταψηφίζουμε όλους τους συμβιβασμούς. Περιμένω Μάλλον θεωρώ ότι στους τελικούς συμβασμούς οι προφορικές δεν θα γίνουν αποδεκτές, αν και μπορούν να υποβληθούν και εγώ θα το κάνω αυτό, για να ε, γίνουμε ε, για να γίνουν ορισμένες ε, διορθώσεις, ιδιαίτερα για την συμπερίληψη των χωρών της περιοχής του Σαχέλ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για ασφάλεια, σταθερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, μέσα στα πλαίσια της ε, UCAP να βελτιώσει την κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ, συμπεριλαμβάνοντας και τη χώρα του Νίγηρα. Είναι ένας ε, τομέας όπου μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και ελπίζω η έκθεση να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, μιλήσουμε με μία φωνή για την κατάσταση της ε, Δυτικής Σαχάρας, τότε θα μπορέσουμε κατά την άποψή μου να επιτύχουμε για τη σταθερότητα, ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την ε, εξαιρετική αυτή εργασία την εργασία του μαζί με τους συνεργάτες. Ε, μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψει την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο και φτάσαμε σε τροπολογία συμβάσμου. Όμως αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας ε, είναι ύψης της σημασίας και τονίζουμε σε μια περιοχή, τονίζουμε μια περιοχή η οποία είναι απομονωμένη. Πρόκειται για πέντε χώρες, 65 εκατομμυρίων ε, κατοίκων. Μιλάμε για δύο εκατομμύρια παιδιά τα οποία πλήττονται από το λοιμό και γι' αυτό θα πρέπει να ε, προβάλλουμε την κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ, διότι πρόκειται για μια ε, περιοχή που γνωρίζει μεγάλη αστάθεια. Δυστυχώς πολλά προβλήματα δεν έχουν ληφθεί υπόψη, δεν υπάρχει πρόγραμμα υγείας για τις γυναίκες, δυστυχώς υπάρχουν ακροτηριασμοί των γυναικών και πολλές φορές η χείρα είναι υποχρεωμένη να ε, παντρευτεί τον ε, γαμπρό της. Αυτό ισχύει στη Μαυριτανία, Τσάντ και Μαλή. Τι μπορούμε να πούμε και για την δουλεμπορία που ισχύει στη Μαυριτανία και στον Νίγηρα. Οι συμβασμοί είναι εξαιρετικοί, αλλά έχουμε πολύ δρόμο να ε, διανύσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε άμεσα και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω κι εγώ όμως ε, υπάρχουν πράγματα που δεν ε, κατανοώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν είναι ισόρροπη αυτή η έκθεση και οι τελευταίες δέκα παράγραφοι δεν σχετίζονται με το Σαχέλα αλλά τη Δυτική Σαχάρα. Αυτό με εξέπληξε και μετά παρετήθηκα. Πολλοί θέλησαν να επιβάλλουν το θέμα της ε, Δυτικής Σαχάρας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πλήττονται σε ολόκληρη τη Σαχάρα και όχι μόνο στη Δυτική. Πολλές τροπολογίες ε, διαφωτίζουν την κατάσταση σε αυτή την περιοχή. Επειδή τα σύνορα λοιπόν είναι διάτρητα, η κατάσταση αυτή μεταφέρεται από τη μία χώρα ή τη μία περιοχή στην άλλη. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας ε, έπρεπε να ε, προωθηθεί και στη Γαλλική Γερουσία, όπου διαχωρίσαμε την περιοχή του Σαχέλ από τη Δυτική Σαχάρα. Οι Σκιώδης ε, έκαναν εξαιρετική εργασία, καθώς και εσείς, κύριε Τάνοκ, είχαν υποβληθεί δεχθεί 341 τροπολογίες και φτάσατε σε 41 συμβιβασμούς. Ε, τα καταφέρατε πολύ καλά εκτός από δύο περιπτώσεις. Όπως σας είπα στο Στρασβούργο, δεν μπορώ να δεχτώ τις 32 και 36 και θα ζητήσω από τους αδέλφους του ΕΛΚ να κάνουν το ίδιο. Ο, η τροπολογία 32 μιλά για την αυτοδιάθεση των Σαχαράουι, κάτι το οποίο ε, λαμβάνει υπόψη την αυτονομία του 2007 που είχε προβάλει το βασίλειο του Μαρόκου. Ως προς το, την 36 μιλά για την αλλιευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιοχής ε, του Σαχέλ. Νομίζω ότι αυτή η εμπορική συμφωνία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή τη στιγμή που την χάνει ε, επαναδιαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ισηγητά, χαίρομαι που συνεργαστήκαμε και θα ήθελα να βοηθήσω και το προσωπικό το οποίο ήταν συνεχώς μαζί μας και μας βοήθησε ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε κύριε ε, Ροάτα. Ο κύριος Σαρλάκη. I just heard... Uh, Άκουσα μόλις τα τελευταία, μόλις πρόλαβα τα ε, τελευταία σχόλια σχόλια για την κατάσταση στην περιοχή του Σαχέλ και της ε, Δυτικής Σαχάρας. Ε, δέχομαι ότι η κατάσταση είναι, ότι η έκθεση είναι ικανοποιητική. Θα ήθελα όμως να υποβάλω ορισμένα σχόλια σε σχέση με τη Δυτική Σαχάρα και αυτή την ανισόρροπη σχέση στην έκθεση. Αυτό είναι γεγονός, ε, δεν είναι ε, ιδιαίτερα ισορροπημένη έκθεση, διότι αρχικά ε, μιλούσαμε, θα έπρεπε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με την περιοχή του Σαχέλ, χωρίς τη Δυτική Σαχάρα. Ε, στη συνέχεια λήφθη απόφαση να ενώσουμε τις δύο εκθέσεις σε μία. Η ομάδα μου υποστήριξε την ιδέα να, είχαν παραμείνει ξεχωριστές αυτές οι δύο εκθέσεις και συμφωνώ με τον κύριο Ροάτα που θεωρεί ότι η Δυτική Σαχάρα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής έκθεσης, ιδιαίτερα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θυμάμαι τη θέση του ΕΛΚ, αλλά εάν ελήφθη απόφαση σημαίνει ότι υπήρξε ευρεία συνένεση. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, όμως θα ήθελα να βρούμε το χρόνο να συντάξουμε μια έκθεση που να ασχολείται αποκλειστικά με τη Δυτική Σαχάρα. Επίσης ε, εκτιμώ το πνεύμα συνεργασίας που ε, δίπε τις ε, συζητήσεις για τους συμβιβασμούς. Ο κύριος Τάνοκ είναι ένας πολύ καλός ισορροπιστής με ε, ιδιαίτερα η στάση του κυρίου Ροάτα ε, που ακριβώς αναφέρει ότι δεν θέλει πια να δεχτεί τις 32 και 36 διότι χάσαμε ένα ολόκληρο πρωινό με τις τροπολογίες συμβιβασμού και θεωρούσα ότι η θέση του ΕΛΚ είχε, ήταν τελική, είχε αποφασιστεί και δεν είχα ακούσει αντιρρήσεις κατά τη συνάντηση εκείνη για τα δύο ζητήματα ζωτικής σημασίας ως προς την ε, αυτονομία, την αυτο, αυτοδιάθεση και την αλλιευτική συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει καταγράφω τη θέση του ΕΛΚ. Όλοι γνωρίζουμε, γνωρίζετε ότι η σοσιαλιστική ομάδα πάντα υποστήριζε και θα υποστηρίζει την αυτοδιάθεση των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρας. Δεν δεχόμαστε τη στάση του Μαρόκου για την αυτονομία των νοτίων περιφερειών και διοικητικών διαμερισμάτων. Αυτό το κάνει για λόγους καθαρά κολυσιεργίας και για λόγους σκοπιμότητας διότι μιλάμε για δικαίωμα αυτοδιάθεσης αυτού του λαού με βάση όλα όσα έχουν αναγνωριστεί από διεθνείς οργανισμούς, αρχίζοντας ε, από τα Ηνωμένα Έθνη και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πάντα υποστήριζε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Δυτικής Σαχάρας και αυτή θα είναι η πάγια θέση των σοσιαλιστών ως προς την αληφτική συμφωνία. Από όσο γνωρίζω, το Κοινοβούλιο έλαβε σαφή θέση με την ψηφοφορία πέρσι. Είχαμε πάνω από 100 ψήφους ε, υπέρ υπέρ της ε, ε, διαγραφής μιας συμφωνίας, απαλυφίες μιας συμφωνίας που είναι άδικη και κατά και αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο. Εάν το ΕΛΚ κρατήσει αυτή τη θέση θα δούμε στο Στρασβούργο κατά πόσο το Κοινοβούλιο θα δείξει την, θα προβάλλει την ίδια στεναρή στάση. Τροπολογία Συμβασμού 41. Εάν άλλοι αποσύρονται, τότε εμείς θα αποσυρθούμε, δεν θα δεχτούμε τη 41. Γιατί υπάρχει αμφισημία ως προς το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Άρα και εμείς θα αποσύρουμε την υποστήριξη της 41. Κύρια Βέμπερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την εξαιρετική εργασία και αυτό το λέω όχι για να είμαι φιλική, αλλά γιατί πιστεύω ότι τα κατάφερε πολύ καλά από δύο απόψεις. ως προς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η απόφαση λήφθη, μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρωτίστως στην περιοχή του Σαχέλ και, από αυτή, υπό αυτή την έννοια ο εισηγητής ε, τόνισε τα βασικά στοιχεία μίζωνος σημασίας που δεν εντάσσονται στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτά που προβάλλει είναι πολύ σωστά και βεβαίως υπάρχουν και τροπολογίες που σχετίζονται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Σαχέλ. Βεβαίως το θέμα της ε, Δυτικής Σαχάρας ε, ε, οδήγησε σε αντιγνωμίες διότι ε, υπάρχουν ε, στενα, υπάρχει στεναρή θέση και στάση και από τους μεν και από τους δε. Υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων. Όμως νομίζω ότι φτάσαμε σε τροπολογίες συμβιβασμού που δείχνουν ότι ο εισηγητής μπορεί και θα ήθελε να δεχθεί ή την υποστήριξη της ε, πλειοψηφίας των βουλευτών. Ορισμένες προτάσεις συμβασμού ήταν πολύ δύσκολες. Είχαμε διαβουλεύσεις μετά από την αρχική συνάντηση, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, και ανέκυψαν και άλλα στο μεταξύ. Η την υποστήριξη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Ορισμένε προτάσεις συμβασμού ήταν πολύ δύσκολες. Είχαμε διαβουλεύσεις μετά από την αρχική συνάντηση, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Και ανέκυψαν και άλλα στο μεταξύ. Η ομάδα μας, η φιλελεύθερη, θέλησαν να υποστηρίξουν στεναρά τις προτάσεις συμβιβασμού, αλλά και εμείς θα αποσύρουμε την υποστήριξη στην 36, γιατί θελήσαμε συμβιβασμό χωρίς την τελική πρόταση για ξεχωριστή ψηφοφορία. Μας ελέγχεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν σε μια πρόταση συμβιβασμού, άρα θα πρέπει να αποσύρουμε την υποστήριξή μας και στη συνέχεια κάθε τροπολογία θα ψηφιστεί ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε την ε, έκβαση της ε, ψηφοφορίας γιατί υπάρχουν ε, πολλές αντιγνωμίες. Είναι πολύ κρίμα. Θα πρέπει να αποστείλουμε ένα μήνυμα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν λέω ότι υπάρχει ομοφωνία, αλλά τουλάχιστον ένα συνενετικό πλαίσιο, αλλά εφόσον δεν είναι δυνατόν, δεν έχουμε παρά να δούμε πού θα μας οδηγήσει η ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε και θα δούμε τι θα συμβεί και στην Ολομέλη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νέλσον, παρακαλώ. Voilà. Oui, merci. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω και εγώ όπως και οι συνάδελφοι ότι δουλέψαμε πάρα πολύ καλά με τον κύριο Τάνοκ, λέει η κυρία Κερνίνσεν, και ο κύριος Τάνοκ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ε, έδειξαν μεγάλη προθυμία και στο Στρασβούργο μάλιστα προσθέσαμε και συνεδριάσεις για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και πολύ με ικανοποιεί ε, η έκθεσή του γενικά επίσης με βρίσκει σύμφωνη και χαίρομαι που μπήκε ένα σημείο που θεωρούσαμε σημαντικό και στην αρχή δεν είχε μπει ε, για ε, την δουλεία λόγω καταγωγής. Δυστυχώς τα θέματα της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών δεν συμπεριλήφθη. Κρίμα, εγώ είμαι πολύ δραστήρια στην Επιτροπή Γυναικών και εν πάση περιπτώσει τι να κάνουμε οι συγητές και οι σκιώδεις ε, έδειξαν προθυμία να συμφωνήσουν ε, οι πολιτικές ομάδες και πραγματικά ευχαριστώ τον κύριο Τάνοκ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε όλη αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα μόνο να πω το εξή χωρίς να επαναλάβω τα όσα είπε ο συνάδελφος Αρλάκη, γιατί η ομάδα μου συμφωνεί για την αυτοδιάθεση της Δυτικής Σαχάρας και του λαού τη και ε, για την αλληλευτική συμφωνία συμφωνούμε και εμείς οι πράσινοι ε, έχουμε την ίδια θέση με τους σοσιαλιστές για τη Δυτική Σαχάρα. Σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ξεχωριστή έκθεση, αλλά μου αρέσει και αυτή τώρα. Γιατί όχι, μια νέα έκθεση αποκλειστικά ε, για τη Δυτική Σαχάρα. Διότι ακριβώς το μεγαλύτερο τμήμα της έκθεσης αφορά το Σαχέλ στο σύνολό του και είναι φυσιολογικό και επόμενο, γιατί αυτό είναι και ο τίτλος, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο η Δυτική Σαχάρα. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πάρα πολλά θέματα και δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνούς δικαίου και πάει λέγοντας. Ε, θα μπορούσαμε και στο μέλλον να κάνουμε νέα έκθεση για τη Δυτική Σαχάρα. Ε, προς το παρόν τώρα έχουμε αυτή, τι να κάνουμε... Έγινε πολλή δουλειά, είναι καλή δουλειά, δεν ήταν καθόλου εύκολο και με βρίσκει ικανοποιημένη η πρόταση. Για τη συμβαστική 41 θα ήθελα να προτείνω μια προφορική και σας το ανακοινώνω από τώρα. Αυτά είχα να προσθέσω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σόλτς παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σκιώδης ηγητές ε, Βίλι Μαγερ και Μαρή Κριστίν Βερζιά κολλείονται και απουσιάζουν και ε, μου ανέθεσαν να σας ε, παρουσιάσω κάποιες παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε, για ένα θέμα δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και ε, έχουμε βοηθήσει και εμείς στις προσπάθειες συνεννόησης. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να προσπαθήσουν να καταλάβουν ε, το συμβιβασμό. Ε, να παραμείνει παρακαλώ αυτή η πρόταση για την αυτοδιάθεση της Δυτικής Σαχάρας. Ξέρετε ποια είναι το ιστορικό αυτής της έκθεσης. Ήταν και μακρύ. Σαχέλ, ε, Δυτική Σαχάρα, χωριστή, όχι ξεχωριστή. Τα ξέρετε αυτά, να μην τα επαναλάβω. Πρέπει πολύ συγκεκριμένα να αναφέρουμε την άποψή μας και να λέμε τι ισχύει. Να σας δώσω τρία παραδείγματα. Για να επανέλθουμε στην ακριβή διατύπωση, ιδιαίτερα στην παράγραφο H, στην αρχική διατύπωση, γιατί είναι και αυτή η διεθνής διατύπωση. Και βέβαια τα Ηνωμένα Έθνη ε, στο ψήφισμα της 11ης Νοεμβρίου του 1980 έχουν εκφράσει ε, την ε, διαμαρτυρία τους για ε, την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα και την κατοχή εκεί. Το ίδιο ισχύει. Και για τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Αναγνωρίζει ότι ούτε το Μαρόκο ούτε άλλοι έχουν ε, αναγνωρίσει ε, τη διοικητική, ε, μάλλον τη δικαιοδοσία του Μαρόκου σε αυτή την περιφέρεια. Θα πρέπει να παραμένουμε στη διατύπωση των διεθνών οργανισμών, εν Όσοι ζητούν να υπάρξει ξεχωριστή έκθεση για τη Δυτική Σαχάρα, βρίσκουν σύμφωνα, είναι πολύ καλή ιδέα και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και έχει αυτή τη δυνατότητα η Επιτροπή μας, αλλά το συντομότερο χρειάζεται άλλη έκθεση. Η κυρία Νέιτς, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τον συνάδελφο Τάνοκ. Συχνά διαφωνούμε με τον κύριο Τάνοκ, οι δυο μας εννοώ, αλλά ε, ε, προκειμένου θέλω να καλωσορίσω και να χαιρετήσω και την ποιότητα της δουλειάς του, γιατί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πέντε χώρες Αχέλη είναι πάρα πολύ περίπλοκη και δύσκολη γενικότερα. Και το θέμα της Δυτικής Σαχάρας ακόμα περισσότερο, όπως φάνηκε και από τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Δεν θέλω να υπάρξει καμία παρεξήγηση, εκτιμώ βαθύτατα ε, το έργο και την προσπάθεια του συναδέλφου Τάνουκ που ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα, θα μιλήσω λίγα λεπτά, όχι πάρα πολλά, ε, κυρίως για τη Δυτική Σαχάρα. Πολλοί ε, από εσά γνωρίζετε ότι γνωρίζω πολύ καλά το Μαρόκο μου, είναι οικία η χώρα και η κατάσταση γενικότερα. Αυτό που έχει σημασία και το βλέπουμε και στην έκθεση είναι ότι επιμένουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτή τη σύραξη. Γιατί διένεξη υπάρχει, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Και θα πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Αυτό που επίσης γνωρίζουμε, και αν θυμάμαι καλά, εμπαρόδο μόνο ε, αναφέρεται ακροθυγός η έκθεση, δεν ε, ενέχεται εκεί μόνο το Μαρακό και τουλάχιστον άλλη μια τρίτη χώρα ενέχεται, που είναι η Αλγερία. Ξέρω ότι ορισμένοι θα διαφωνήσουν και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της από την αρχή, έτσι ώστε να ε, εμποδίσει τη λύση. Μια ενδεχόμενη προσέγγιση για να φτάσουμε σε μια λύση είναι ο σεβασμός των γεγονότων. Πρώτο, σε μία από ε, τις συμβιβαστικές γίνεται λόγος για 13 θύματα κατά την εκένωση του προσωρινού καταβλισμού στη Δυτική Σαχάρα. Δεν λέγεται όμως ότι και τα 13 θύματα είναι μέλη των Μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας. Ήταν αστυνομικοί οι οποίοι κυριολεκτικά κατακρεουργήθηκαν. Είναι γεγονότα αυτά, δεν επινοώ τίποτα. Ε, όταν στη συμβιβαστική 36 αναφέρουμε ότι το κοινοβούλιο μας ε, απέριψε την προσωρινή αλληλευτική συμφωνία, αυτό με ενισχύει πλην όμως. Δεν ήταν ξεκάθαρο τι γίνεται με τα κέρδη από αυτή την αλία. Ότι ε, δεν ήταν ξεκαθαρισμένο ότι θα πήγαιναν τα κέρδη ε, στο λαό Σαχράουι, αλλά δεν ήταν ο μόνος λόγος απόρριψης. Εγώ συμμετείχα στην ομάδα μου στη συζήτηση, παρακολούθησα τις εργασίες και μεταξύ άλλων η Επιτροπή αλλιές ήταν ε, πολύ λίγο ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο απάντησε ή δεν απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης το γεγονός ότι Εκάλυπτε μια χρονιά αυτή η συμφωνία από την οποία ε, το μόνο τέσσερις εβδομάδες. Οπότε είπαμε στην απορρίψουμε τι θέλουμε. Και με βάση αυτό να συστήσουμε στην έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο να απορρίψει μια αλληλευτική συμφωνία που είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης και που ακόμα δεν γνωρίζουμε την έκβαση Αυτή είναι κάτι που εγώ δεν μπορώ να δεχθώ. Και γι' αυτό το λόγο εμείς αποσυρθήκαμε από το συμβιβασμό και είναι πολύ σημαντικό πρώτα να κάνουμε εμεί τον εαυτό μα συστάσει για ένα κείμενο το οποίο γνωρούμε. ε, πώς να το πω, είναι λίγο παράτολμο. Ε, τέλος θα ήθελα να συγχαρώ όχι μόνο τον Τσάλ τάνοκ που κάνει καταπληκτική δουλειά, αλλά όλους τους ε, εισηγητές μας, τους σκιώδεις όπως ονομάζονται, γιατί όλες οι ομάδες μας είναι διχασμένες σε αυτό το θέμα. Και οι σκιώδης ηγητές χρειάζεται και να επιδείξουν ε, και διπλωματία αλλά και επιδεξιότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό και τη γραμματεία της ε, Επιτροπής αλλά και τους βοηθούς των ομάδων μας. Μου κάνει πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παντζέρη, παρακαλώ. Grazie Presidente, mi associo anch'io a Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ και χειροκροτώ τον κύριο Τάνοκ. Πολύ καλή μου φαίνεται η έκθεση αυτή. Και όταν μιλούμε για το Σαχέλ και τα προβλήματα ε, που γνωρίζει, υπάρχουν βασικά ζητήματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα που συνδυάζονται και με ευρύτερα προβλήματα ασφαλείας, γενικότερα περιφερειακά, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που έχουν τα ζητήματα ασφαλείας και στις υπόλοιπες χώρες και κατά συνέπεια και ε, στην Ευρώπη. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα λίγο να σταθώ στη Δυτική Σαχάρα. Θα προσπαθήσω να εκφράσω μία άποψη και να απαντήσω λίγο στα όσα μόλις άκουσα πριν ψηφίσουμε στην Ολομέλεια, ο καθένας από εμάς θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει στην ομάδα του αυτό το θέμα. Δεν θα κάνω μια κρίση, μια γενική παρατήρηση μόνο. Για το θέμα αυτό δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφραστεί. Η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε εμπλοκή μεταξύ εκείνων που θέλουν την αυτοδιάθεση και εκείνων που θεωρούν ότι αποκλείεται και ότι είναι ανέφικτος αυτός ο στόχος. Νομίζω ότι θα έχουμε απροσπέλαστες δυσκολίες σε σχέση με τις αρχικές μας θέσεις. Τη στιγμή που επί δεκαετίες δεν έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών τη στιγμή που δεν έχουν γίνει ουσιαστικά ε, και ορατά βήματα προς τα εμπρός. Θεωρώ και εγώ ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη θέση του Μαρόκου και της Αλγερίας. Και ίσως θα ήταν σκόπιμο, αν θέλουμε να συνεισφέρουμε πραγματικά, και να μην προβαίνουμε σε διελκυστίνδες, να ενισχύσουμε αυτή την ιστορική φάση βρίσκοντας ε, λύσεις με μικρά βήματα σε σχέση με την ε, τελική στοχοθέτηση. Αυτό θα ήταν επιθυμητό. Βεβαίως χρειάζεται ε, θάρρος, μεγάλη προσπάθεια και όχι μόνο φαντασία σχετικά ως προς την αρχική μας θέση αυτών που τάσσονται υπέρ και εκείνων που τάσσονται κατά. Γιατί νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις συμβιβασμού δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν στην ε, τελική ψηφοφορία και δεν θα έχουμε υπηρετήσει ε, μια τέτοια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή της Δυτικής Σαχάρας. Μίλαν μόνο. Ευχαριστώ εντάχει. Δεν ξέρω αυτές τις τροπολογίες συμβιβασμού της επίπονες που έτυχαν διαπραγμάτευση υπό, υπό τον κύριο Τάνοκ. Είναι 41 νομίζω. Ως προς τη 36 τώρα θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου σε σχέση με την αλληλευτική συμφωνία με το Μαρόκο. Εγώ ήμουν πέρ της διατήρησης αυτής της συμφωνίας αρχικά πριν από δύο χρόνια. Εμείς είμαστε υπέρμαχοι αυτές, αυτής της αλληλευτικής συμφωνίας, η οποία είναι ευεργετική και για, τους ευρωπαϊκούς, για τον ευρωπαϊκό ε, στόλο. Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ε, περιοχή του Σαχέλ και της Δυτικής Σαχάρας και δεν, μιλάτε, δεν γίνεται λόγος για την αλληλευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου. Και με βάση τον τίτλο της έκθεσης δεν μπορούμε να μιλάμε αποκλειστικά για ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί υπάρχουν και πολλοί Σαχαράουι οι οποίοι επανδρώνουν αυτό το, το στόλο, τον ε, μαρακινό στόλο. Ο κύριος Σαρλάκη, εντάχει όμως σας παρακαλώ. Ο κύριος Σαρλάκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση. Ε, ανέφερε η κυρία Νέιτς ένα ατύχημα, που, μια ατυχή, ένα ατυχές συμβάν που είχε να κάνει με την μαροκινή αστυνομία, αστυνομικές δυνάμεις, αλλά υπάρχει μια διαφορετική εκδοχή, την οποία θεωρώ πιο αξιόπιστη, ότι 80 αρχάου είχαν φωνευθεί κατά τις συγκρούσεις με ε, την αστυνομία και η δίκη ήταν τελείως άδικη, διότι κάθε στοιχείο αποδεκτικό το οποίο θα οδηγούσε σε καταδίκη ή θα μπορούσε να επιρρύψει ευθύνε στην αστυνομία της, ε, από τους αστυνομικούς από το Μαρόκο, απερίφθη και δεν ελήφθη υπόψη. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε καταστάσεις. Πολίτες διαδηλώνουν παρεμβαίνει ένοπλη αστυνομία μαροκινή με πολύ σκληρή καταστολή και μετά καταδικάζονται οι λεγόμενοι προτεργάτες, υποκινητές των διαδηλώσεων. Ο κύριος Παντζέρη επίση αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η διεκδίκηση για αυτοδιάθεση, αν δεν επιτυγχάνεται, πρέπει να αλλάζει ή να αποσύρεται. Απαράδεκτο αυτό. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα πρέπει οι Παλαιστίνοι να παραδεχθούν την ε, κατοχή ε, του Ισραήλ, γιατί η κατάσταση δεν προχωράει, ή σε όποιο άλλο κράτος διεκδικούνται το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και άλλα δικαιώματα, θα πρέπει να υποχωρούν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν τον αγώνα. Αυτό είναι ο λόγο νομίζω για τον οποίο όλε οι διεθνεί οργανώσει, διεθνέ δικαστήριο, Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεξή και ούτω καθεξή αναμφίβολα και απερίφραστα και απεριόριστα υποστηρίζουν τα άνθρωπινα δικαιώματα. Η κυρία Νέτση έχει το λόγο. Στα γαλλικά. Πολύ σύντομα, πρόεδρε. Καταρχάς, ούτε και θα μου παίρναγε από το μυαλό να αποτελέσω ατυχές συμβάντα όσα συνέβησαν σε αυτό το ε, καταβλισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσα συνέβησαν, συνέβησαν με ε, στρατιωτικά, μέσα, σύμφωνα και με το Σύνταγμα του Μαρόκου την εποχή εκείνη. Επιτρέψτε μου να ομιλήσω, σας παρακαλώ. Ότι πολλές από τις δικές μας χώρες, μέχρι ακόμα λίγο χρονικό διάστημα, ε, επίσης περνούσαν από στρατοδικείο τέτοιου είδους υποθέσεις. τελευταίες δεκαετίες μόνο άλλαξε σχετική νομοθεσία. Είναι δημόσια η δίκη, ήταν δημόσια και την παρακολούθησαν και μέλη της ε, Μαροκινής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αλλά και διεθνείς παρατηρητές οι οποίοι διακήρυξαν γενικά την ικανοποίησή τους για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η δίκη αυτή. Άλλωστε εγώ τους έχω μιλήσει προσωπικώς και με την Αντιπρόεδρο της Οργάνωσης των τα Ανθρωπινά του Μαρόκου. Επίσης, η κυβέρνηση του Μαρόκου απεφάσισε και άλλαξε τον νόμο ώστε να μην παραπέμπονται πλέον σε στρατοδικείο τέτοιου είδους περιστατικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε το υπογραμμίσαμε και στην ε, συμβαστική μας πρόταση. Κύριο Σπάσκου, Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι και ο κύριος Παντσέρη θα στο λόγο τώρα, αλλά θα παρακαλέσω τους πάντες να μην ξαναρχίσει αυτή η συζήτηση, να μην γίνει μια συζήτηση μέσα στη συζήτηση. Κύριε Παντσέρη. Εάν δεν μου επιτρέπετε ανταπάντηση, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί ένας διάλογος. Δεν πρέπει να συγχαίουμε το νομικό πλαίσιο που τη στιγμή που έχει οριστεί και πρέπει να τηρηθεί από την πολιτική διαδικασία. Γιατί διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από την εκτέλεση του νόμου. Αλλά εμείς είμαστε ένα κοινοβούλιο και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πολιτικά βήματα που θα μπορούσαν να προωθηθούν για να φτάσουμε στο στόχο μας. Έχουμε υποχρέωση να μιλήσουμε για αυτά τα πολιτικά βήματα, γιατί τότε δεν έχει νόημα ούτε καν να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει από τα Ηνωμένα Έθνη, άρα δεν έχουμε παρά να παραμείνουμε εκεί. Εάν θέλουμε όμως να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, θα πρέπει να δεχτούμε την άποψη όλων. Διαφορετικά παραμένουμε στάσιμοι στις αρχικές θέσεις και θα δούμε πώς θα επιληθεί το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σε ΙΕΔ, ο κύριος Περνάς Σαλβάζ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να επαναλάβω τη σημασία ε, του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις ε, δράσεις της ΕΙΕΔ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα με τρίτες χώρες. Όμως, θα πρέπει να σχολιάσουμε ορισμένες πτυχές του, της τροπολογίας Συμβασμού 36 σε σχέση με την παράγραφο 40. Πρώτον, σε σχέση με την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών που παρατίθεται. Η προηγούμενη παράγραφος αναφέρεται και στην 25 Εάν υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη παρά τη θέληση της Δυτικής Σαχάρας, τότε παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο σε σχέση με τους ορικτούς πόρους της περιοχής αυτής. Άρα η νομική θέση δεν εξαιρεί την εκμετάλλευση του ορικού, ορυκτού πλούτου. Η Συμφωνία Σύνδεσης και η Συμφωνία για τη Γεωργία και την Αλία αφορούν και το Βασίλειο του Μαρόκου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχετικές ε, δηλώσεις της 16 Φεβρουαρίου του 12 σε σχέση με την εμπορική συμφωνία στο εμπόριο και τη γεωργία θεωρεί ότι το Μαρόκο θα πρέπει να ανταποκριθεί ως προς τον αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας. Έχουν οριστεί οι, τρόποι ε, επικοινωνίας. Η πρώτη Τη αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη θα γίνει στην περιοχή τον επόμενο μήνα. Το ίδιο αφορά και το αλευτικό πρωτόκολλο της 30 Σεπτεμβρίου του 2011. Δεν μιλάμε μόνο για την κάλυψη της Δυτικής Σαχάρας καθεαυτής, αλλά για τους όρους εφαρμογής αυτού του πρωτοκόλου. Στη Δυτική Σαχάρα το Κοινοβούλιο ζήτησε μια εκτενή έκθεση όλων των δραστηριοτήτων δυνάμει αυτού του μελλοντικού πρωτοκόλου. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα προβληματικό στοιχείο στα συμπεράσματα μέσα στο συμβιβασμό, που υπάρχει στο συμβασμό 36, σε σχέση με την αιρεσιμότητα, διότι εδώ δεν πληρούνται οι όροι. Και θεωρείται ότι η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου δεν λαμβάνει υπόψη τα, τις επιθυμίες ε, της ε, περιοχής της Δυτικής ε, Σαχάρας. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάθε εκμετάλλευση και οι σχετικές διακλαδώσεις της συμφωνίας αυτής παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Νομίζω ότι κινούμαστε γύρω-γύρω κυκλικά στην υπόθεση αυτή, δεν καταλήγουμε πουθενά αυτή. Θα αντιλαμβάνεστε γιατί ήταν τόσο δύσκολη αυτή η έκθεση, από τις πιο δύσκολες τα 14 χρόνια που στο Κοινοβούλιο. Αλλά πάντως η υποεπιτροπή των ανθρωπινών δικαιωμάτων ε, ήταν αυτή η οποία ανέλαβε την έκθεση και όχι άφετ για τις μέρους παρεμβάσεις των συναδέλφων, σκιωδών, συγκεκριτών και άλλων. Τον κύριο Ρώτα, θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ ότι ε, παραμελήθηκε τα δικαιώματα στην υγεία των γυναικών. Εγώ δεν θα ήθελα τον όρο αναπαραγωγική, όπως θέλει η κυρία Κινίλσον, γιατί ουσιαστικά πίσω από αυτό υποκρύπτεται η άμβλωση. Πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με τι πεπιθήσει μου περί ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όποιο θέλει να το συμπληρώσει, εγώ δεν θέλω να το βάλω στην έκθεση με το δικό μου χέρι. Στα άλλα θέματα. Ε, καταναγκαστική γάμη είναι ζητήματα τα οποία είναι πολλές φορές ιδιαίτερα ή χαρακτηριστικά μίας ε, χώρας ε, για την για τους όρους που έχουμε στα αγγλικά, άλλωστε χρειάζεται κανείς να ανατρέξει στο λεξικό για να καταλάβει, στο θέμα της ε, δουλείας φαίνεται ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει στην περιοχή. Δυτική Σαχάρα. Είπατε ότι θέλετε το 32 και το 36 να προσεχθούν. Εγώ δεν θέλω να είμαι πολύ απόλυτος και μεροληπτικός ως προς το ενδεχόμενο μιας λύσης του ζητήματος και την αναφορά το εις αρχής της αυτοδιάθεσης ή της αδαφικής ακαιρεότητας. Παραμένω ε, επί τούτου αμφίσιμος γενικόλογος στην τοποθέτησή μου για να μην τοποθετηθώ και κατηγορηθώ ότι μεροληπτώ. Η αλία είναι ένα ζήτημα καυτό στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μιλανμόν ομολογεί ότι οι Ισπανοί έχουν μέγα συμφέρον στην αλία. Οι Ισπανοί ούτως ή άλλως έχουν εδώ και 40 χρόνια αποτραβηχθεί, έχουν υποχωρήσει, έχουν μάλλον ε, απεμπλακεί από την υπόθεση αυτή. Και όπως είπε και ο κύριος υπάρχει μια εκδηλώθηκε μάλλον μια ευρεία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την απόρριψη της συμφωνίας, ε, αλληλευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο. Αν και με τη δική μου διατύπωση δεν αποκλείεται η εκμετάλλευση των πόρων στο βαθμό που είναι προς το συμφέρον των ε, κατοίκων. Δεν είμαι νομικός, εάν η νομική μας ε, υπηρεσία θεωρεί ότι είναι αντίθετο με τους κανόνες του δικαίου αυτό που γράφω, ας μας διορθώσουν. Κύριο Σαλάκη επιδιωκεί αντίστοιχους στόχους φαντάζομαι αλλά με διαφορετική προοπτική, άρθρο 36-41. Κυρία Βέμπερ, λυπούμε που αποσύρει την υπογραφή της η από το 32 και σε έναν παραγωγική για το ε, ε το έδειξα, το κάλυψα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για έκθεση σχετική με το διεθνέ δίκαιο. Είναι μια έκθεση σχετική με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Φυσικά έχει σημεία επικάλυψης ε, αρκετά με το Δημόσιο Δίκαιο. Κυρία Νέιτς, ναι, όντως ευαίσθητο θέμα, συμφωνώ. Χωρίς όμως να είναι στόχος της εκθέσεώς μου να επιλύσω ή να, βρω, να δώσω απαντήσει αυτή την ε, ε, χρονίζουσα σύγκρουση. Ίσως στο 34 θα μπορούσε, αν θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο, να ενσωματωθεί η τροπολογία σας για την ε, αναφορά των ονομάτων των 13 θυμάτων. Ε, ο κύριος Παντσέρη γνωρίζει ασφαλώς περισσότερα από ότι εγώ στην, ε, για την περιοχή αυτή, αλλά θα συμφωνήσω εγώ με τον κύριο αλλά και ότι δεν μπορεί η αυτοδιάθεση να διαγραφεί ή να απεμποληθεί όταν δεν καθίσατε αμέσως εφικτή. Υπάρχουν βέβαια και άλλες λύσεις, αλλά θα πρέπει να είναι αποδεκτές για τις δύο πλευρές, για κάθε πλευρά και με μια παραπομπή στην παρθενική μου ομιλία για το Ανατολικό Τιμόρ πριν από 14 χρόνια εδώ, θα ήθελα να πω ότι αν δεν είχαμε καταλήξει τι προσπαθίε με γιατί φαίνεται ορατή αυτοδιάθεση του ανατολικού Τιμόρ, θα ήταν τελείω διαφορετική η κατάσταση στην Ινδονησία. Το ίδιο θα ίσχυε και για, την, για πολλές χώρες Αφρικής, Ναμίβιο και το καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει κάθε αγώνας για αυτοδιάθεση, κάθε λαός που αγωνίζεται για την αυτοδιάθεσή του να αξιολογείται και με βάση τις πράξεις του στο δημόσιο διεθνέ δίκαιο και αναλόγως να κρίνεται η κατάσταση. Δεν βλέπω να μιλάει κανείς για το υπόλοιπο Σαχέλ πριν τη Δυτική Σαχάρα από όσου μίλησαν. Αλλά για να επανέλθω στο κύριο ζήτημα, κύριε Αλάκη... Νομίζω ότι ε, έχετε λάθος ε, πληροφορίες και εγώ άλλωστε είχα ενημερωθεί σφαλμένα στην αρχή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τη δική Σαχάρα, ένα, ένα μια πρόταση που ξεκίνησε από τη δική σας την ομάδα. Εγώ όταν ε, είχε ήδη μετα, μετονομαστεί και μετατραπεί σε Συμφωνία Σαχέλ είδα το θέμα και το ανέλαβα. Μετά πρόταση στον κύριο Μπροκ ζητούσε να μετατραπεί, να διευρυνθεί στην, στην, ε, στο ζήτημα όλης της Σαχάρας. Επανήλθαμε στο Σαχέλ, εν πάση περιπτώσει. Όπως είπα, γυρνάμε γύρω-γύρω. Ξεκινήσαμε από τη Δυτική Σαχάρα. Και όποιος θέλει να αναλάβει έκθεση για τη Δυτική Σαχάρα, με γεια του, με χαρά του και καλή δύναμη, αλλά θα σας ε, προειδοποιήσω ότι είναι πολλά τα λόμπι, οι πιέσει και οι δυσκολίες στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ολοκληρώνουμε έτσι τη συζήτηση. Το επόμενο θέμα στη μέση Ένταξη. Θα διευκρινίσω κάτι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Γκόμες. The So, για τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν αντί αυτής της διατύπωσης, ενώ παραμένει ανεπίλητη αυτή η διένεξη, δηλαδή που παραπέμπει στην όλη σύγκρουση, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ενώ οι αναφορές που μαθαίνουμε και οι ειδήσει ε, δεν θεωρούνται ικανοποιητικέ ε, σύμφωνα με το λαό της Δυτικής Σαχάρας, το Σαχράου. Εντάξει, θα το δω αυτή τη διατύπωση με τις νομικές μας υπηρεσίες, εκπρόσωπος. Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με τον δόκτωρα Σίμα Σάμι Μπαούς, Διευθύντου του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τι Αραβικέ χώρε. Την κυρία Μπαούς. Κατόπιν μιας υποδηματική σταδιοδρομία στην Ιορδανία, η κυρία Μπάχους, η δόκτωρ Μπάχους, έχει αναλάβει την ε, διεύθυνση 18 ε, γραφείων αντιπροσωπιών σε αραβικές χώρες τον, ε, του προγράμματος ανάπτυξης των Εθνών. Θα θέλαμε βεβαίως να ακούσουμε τι συμβαίνει στη Συρία και τι είδους επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κατάσταση για τις γειτονικές χώρες. Μα απασχολεί το θέμα, το έχουμε ξανασυστήσει. Θέλουμε να ακούσουμε τις δικέ σας απόψεις και εκτιμήσεις και συστάσεις. Άλλε σημαντικές χώρες όπως η Αιγύπτος, η Τινησία, η Λιβύη ακόμη δεν έχουν ε, γνωρίσει την ειρήνη και την ηρεμία. Μια σειρά από προβλήματα λοιπόν ε, επικρατούν στις χώρες αυτές και αναπόφευκτα συνδυάζονται κιόλα μεταξύ τους για να επιδεινώσουν την κατάσταση. Θα σα παρακαλέσω να λάβετε το λόγο για περίπου 10 λεπτά για να προχωρήσουμε μετά σε διάλογο με τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάσου. εξωτερικοί κυρίε και κύριοι του Κοινοβουλίου. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ Προέρχομαι από μια περιοχή και εκπροσωπώ μια περιοχή που όπως γνωρίζετε γνωρίζει κρίση σήμερα. Ε, εκπροσωπώ και μια ε, η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυξη που καταβάλει κατά δυνατή προσπάθεια, αναζητώντα ε, τρόπου για την δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όπω γνωρίζετε, πριν από τρία χρόνια ανέλαβαν ε, θαραλέα βήματα στο μεγάλο δρόμο για τη δημοκρατία οι, λαοί, οι αραβικοί λαοί. Κατέβηκε ο κόσμο στου δρόμου, ζητώντα να διαμορφώσει μόνο του το μέλλον του, απορρίπτοντα ε, την ανεργία, τη φτώχεια, την την ανησυχία για το μέλλον. γυναίκε άντρε και παιδιά κατέβηκαν στον δρόμο για να στήσουν ένα νέο μέλλον που ενέπνευσαν με τον τρόπο αυτόν όλη την περιοχή του, την ευρύτερη περιοχή αλλά και όλο τον κόσμο. Ζητούσαν με την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπειά τους, ε, διεκδικούσαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καλύτερη ποιότητα ζωή. Και φαινόταν ότι αυτό θα μπορούσαν να το επιτύχουν. Τώρα όμω βλέπουμε ότι σβήνουν οι ελπίδες και καταπέφτουν στην απόγνωση αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπουμε την ε, βία, τη, τους αγώνες, τους θανάτους, ε, τις συγκρούσεις στην Ιεμένη, τη Λιβύη, τη Συρία βεβαίως πάνω από όλα τη Συρία στην οποία βλέπουμε να χάνουν τη ζωή τους τόσοι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια να είναι αυτοί που φεύγουν από τις αιστείες τους. Πάνω από 100.000 άνδρες, γυναίκες, παιδιά που ξέρετε έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν, χάσει τις, έχουν φύγει από τις αιστείες τους. Πάνω από 4 εκατομμύρια έχουν φύγει στο ιστορικό της χώρας σε κάποιες άλλες περιοχές. Σχολεία, σπίτια, ε, νοσοκομεία έχουν κατεδαφιστεί η κατάσταση ανθρωπιστική είναι κατεπίγουσα και η μετάβαση, η ανάκαμψη, η ανάπτυξη δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Γι' αυτό λοιπόν πάνω απ' όλα για το μέλλον της Συρίας, της Ίνδιας, αλλά βεβαίως και για τις προοπτικές ε, των όμορων και γειτονικών κρατών, για την υποπεριφέρειά της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί μια λύση στην, ε, στην κρίση αυτή, γιατί πιέζεται ιδιαίτερα όλη η περιοχή, η Ορδανία, ο Λίβανος, πιο πρόσφατα το Ιράκ, που συνταράσσονται από αυτή την κρίση και χρειάζονται την υποστήριξη των διεθνών εταίρων. Οι χώρες ε, υποδοχή στην Ιορδανία και τον Λίβανο αλλά και το Ιράκ πιο πρόσφατα βλέπουν το μεγάλο βάρος της υποδοχής των προσφύγων και της διάθεσης πόρων σε κάθε επίπεδο. Ανά τον αραβικό κόσμο βλέπουμε να επικρατούν δύο οράματα και να αντιπαρατίθενται δύο οράματα. Το ένα που κοιτάει στο μέλλον την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία και τη ελευθερία και το άλλο που είναι η απόγνωση. Το πιο όραμα θα επικρατήσει είναι κατά την άποψή μου, κατά την άποψή σας, κατά την άποψη του Οργανισμού των Εθνών και του Προγράμματος για την Ανάπτυξη, αυτό που θα εξαρτηθεί από την αηφόρο ανάπτυξη, αυτό που θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα χειριστούμε την αηφόρο ανάπτυξη στην περιοχή αυτή, για την τελευταία ανάλυση όλη αυτή η ενώ κατ, κατ' επίφαση ήταν... Ε, αγώνες, ε, στην επιφάνεια του ήταν αγώνες για τη δημοκρατία, κατά βάθο είχαν σαρίζα τον αποκλεισμό, τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό, την απογνώση. Οι θέσει εργασία ε, που ήταν πάρα πολύ περιορισμένε η ανεργία και κυρίως των νέων είχαν επιδεινώσει αυτή την ε, κατάσταση ευαισθησία, αυτή την τόσο ασταθή κατάσταση στι χώρε αυτέ, που τώρα πια έχουν φτάσει σε ορισμένα σημεία να έχουν προβλήματα ακόμη και διατροφικά. Μεγάλοι πληθυσμοί λοιπόν, πολύ η πληθυσμοί και νέων, φτώχεια, εξαθλίωση, Σομαλία, ε, ε, Λιβύη και άλλες περιοχές, όπως ξέρετε, μπορούν να προσφέρουν ε, γόνιμο έδαφος και υλικό ε, ανθρώπινο για τους εξτρεμιστές. Και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Προσπαθούμε να ανατρέψουμε λοιπόν την στασιμότητα και στην ανάπτυξη του αραβικού κόσμου, πράγμα το οποίο αποτελεί μια προϋπόθεση αναπόδραστη για την διασφάλιση του μέλλοντος της περιοχής αυτής. Δεν υπάρχει μετάβαση και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε ιστορικά που να μην έχει προχωρήσει κατά τρόπο που να έχει προχωρήσει κατά τρόπο απρόσκοπτο ή ταχύτατο. Άρα δεν χρειάζεται να απογοητευόμαστε και να πέφτουμε σε απόγνωση. Χρειάζεται η προσπάθεια όμως να συνεχιστεί. Χρειάζεται να κερδίσουμε την υποστήριξη των πολιτών και επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε τα λοιπά χαρακτηριστικά της περιοχής, την, το έλλειμμα γνώσης, το έλλειμμα ισότητας των φύλων για τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια, το έλλειμμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το έλλειμμα κράτους δικαίου και χρηστής διακυβέρνησης. Έτσι λοιπόν πρέπει και τα κράτη αλλά και τους πολίτες να στηρίξουμε για τον, ε, για τον προσδορισμό ενός νέου κοινωνικού συμβολέου, ενώ μιας νέας κοινωνικής σύμβασης η οποία θα βελτιώσει την ποιότητα ζωή, Θα βελτιώσει τη δημοκρατία, θα βελτιώσει, θα βελτιώσει την κατάσταση εν γέννη. Το πρόγραμμα λοιπόν για την ανάπτυξη των εθνών αγωνίζεται με όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε όλες τις αραβικές χώρες όπου υπάρχει ανάγκη για να ρίξουμε τα θεμέλια της ειρήνης και τη δικαιοσύνη, τη ασφάλεια, τη ε, ε, χρηστής διακυβέρνησης, της ε, στη δημόσια ζωή. Αγωνιζόμαστε για να ολοκληρώσουμε το έργο που άφησε ατελείωτο το σύνολο των στόχων για την χιλιετία και να προσδιορίσουμε την, ε, το θεματολόγιο την ανάπτυξη μετά το 2015. Αγωνιζόμαστε επίσης για να στηρίξουμε τις χώρες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας, της, ε, ώστε να δράξουν τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη. Για την Τινησία, παραδείγματι, έχουμε προσφέρει υποστήριξη ουσιαστική και για τις εκλογές και για την διακυβέρνηση και για το κράτος δικαίου. Στην Αίγυπτο εμείς προσφέρουμε προοπτικές και σεβασμό για τα δικαιώματα όλων των πολιτών και καλούμε για ε, στήριξη οικονομική των πιο ευάλωτων. Στη Λιβύη το σύστημά μας, όπως συμπεριλαμβάνεται και το δικό μας πρόγραμμα, προσφέρει ε, στήριξη στις πρώτες ελεύθερες εκλογές στην ε, Λιβύη και ιδιαίτερα προωθεί ε, υποψηφιότητες γυναικών. Υποστηρίζουμε τη θέσπιση του νέου συντάγματος, τη χάραξη πρώτα σύνταξη και θέσπιση του νέου συντάγματος, σε χώρες οι οποίες παίρνουν μέσα από συγκρούσει ή που επηρεάζονται από ενόπλε συγκρούσει σε γειτονικά κράτη. Προσφέρουμε στο βαθμό του δυνατού ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε προγράμματα για τη δημιουργία θέσεων εργασία, διασφάλιση εισοδημάτων και διαφύλαξη τη κοινωνική συνοχή, που με τον τρόπο αυτό μα επιτρέπει να γεφυρώσουμε την ε, ανθρωπιστική βοήθεια με τη μακροπρόθεσμη ε, στήριξη για την ανάπτυξη. Σταθεροποίηση λοιπόν χωρών όπως η Ορδανία και το Μαρόκο, οι οποίες ακόμη δεν έχουν ε, δεν έχουν πέσει, δεν έχουν περιπέσει σε ένοπλη σύγκρουση και ελπίζουμε ότι θα ξεφύγουν από αυτήν, χρειάζονται οπωσδήποτε υποστήριξη για ε, σταθεροποίηση και είναι, είναι ορόσημα στην σταθεροποίηση όλης της περιοχής. Οι αρχές λοιπόν των δικαιωμάτων της δημοκρατίας, στήριξη και εξασφάλιση ευκαιριών για την νεολαία, ε, υποστήριξη της νεολαίας ώστε να βρει τον τρόπο να εκφράσει τη φωνή της, ε, θεματολόγιο για τις γυναίκες. Κοινωνικά και οικονομικά θέματα, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Είναι τα κλειδιά για την επιτυχία στην πολιτική μετάβαση και πρέπει να υπογραμμίσουμε και τη σημασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων και το σεβασμό της, ε, του διαφορετικού και της χρηστής διακυβέρνησης. Εξοχότα ότι με μεγάλη χαρά να πτήσουμε αυτή την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς ε, μας στηρίζουν οι ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθεια αυτή το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών προσπαθεί να προσφέρει αμερόληπτη και ουσιαστική στήριξη και συμβουλές στην περιοχή. Έχουμε μακρά εμπειρία από την ανάπτυξη και ταχύρυθμων προγραμμάτων με ουσιαστικά και γρήγορα αποτελέσματα στις περιοχές ε, της, ε, όπου παρουσιάζονται ενόπλες συγκρούσεις, εμπόλεμες περιοχές. Έχουμε με τα Ηνωμένα Έθνη αναπτύξει αυτή την ε, προσπάθεια και πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε και να παραμένουμε εταίροι του αραβικού κόσμου ακόμη. Είναι άλλωστε ο ευρωπαϊκός κόσμος με τον αραβικό πολύ στενά συνδεδεμένοι. Η αδίποτε επιβράδυνση ε, στην μία ή την άλλη περιφέρεια μπορεί να επηρεάσει ε, τον εταίρο Πολλοί είναι οι νέοι Άραβες οι οποίοι οραματίζονται ευκαιρίες για κατάσταση και εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δικός μας στόχος και όραμα είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι Άραβες, τα 200 εκατομμύρια νέων Αράβων που είναι κάτω από 24 ετών, θα βρουν ε, την ε, θέση τους στη ζωή και, το, και την υλοποίηση των οραμάτων τους στις ίδιες τους πατρίδες. Η ειρήνη λοιπόν, η ειρήνη και η ε, ασφάλεια που κινδυνεύουν και από τους εξτρεμιστές ε, πρέπει να, προστατευθούν, πρέπει αυτό να γίνει μαζί με την ε, υλοποίηση των οραμάτων των Αράβων, των Αραβικών λαών και αυτό βέβαια χρειάζεται και υπομονή και επιμονή και ακαταπώνητες προσπάθειες. Εμείς θα συνεχίσουμε για να κρατήσουμε ζωντανή τη φλόγα της ελπίδας για τους αραβικούς λαούς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, the floor to our... Πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να καλωσορίσω ενώπιόν μας τρία μέλη της Βουλής του Τζιμπουτή, ο κύριος Παΐς, ο κύριος Αμπτιλάχη και ο κύριος Σαΐτ Παρευρίσκονται στις Βρυξέλλες εν ώψη και της νέας συμφωνίας για τη διάσκεψη για τη Σομαλία που διεξήχθη χθε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Παντζέρη, παρακαλώ, και μετά στους υπολείπους συνάδελφους. Sir Robert, and then this is next. Okay. So, Mr. Panzeri. molto, molto brevemente volevo... Εντάχει, θα ήθελα να χαιρετήσω την υπεύθυνη, τη διευθύντρια του προγράμματος και να εκφράσω μία σκέψη και δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η σκέψη μου έχει ως εξής. Συμφωνώ, με όσα προβάλλατε και είμαι όλο ένα και περισσότερο πεπισμένος ότι όσο αφορά ολόκληρη την περιοχή στην οποία αναφερόμαστε θα πρέπει να συνοδεύουμε την δημοκρατική σταθερότητα με μια αναπτυξιακή πολιτική και πολιτική οικονομικής ανάπτυξης, διότι εάν οι άνθρωποι δεν έχουν γεμάτο στομάχι, δεν εκτιμούν εύκολα τη δημοκρατία. Γι' αυτό αυτή η πορεία θα πρέπει να ε, έχει συνοδευτικά μέτρα για την δημοκρατική σταθερότητα της περιοχής και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στη συνέχεια βάλω δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα τη γνώμη σας ως προς την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της πολιτικής More for More διότι πολλοί λένε επί της ουσίας ότι είναι μια ε, σωστή πολιτική, δηλαδή να ε, χορηγούμε όλο και περισσότερα σε εκείνους που κινούνται προς ε, δημοκρατικά καθεστώτα. Άλλοι όμως λένε ότι με αυτή την, σε αυτή την περίπτωση τιμωρούμε τις χώρες οι κυβερνήτες των οποίων δεν μπορούν να προωθήσουν δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο μας απασχολεί εκ νέου. Θα θέλαμε τη δική σας ε, γνώμη για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Δεύτερον, πολλοί αναλυτές λένε το εξή και ξέρω ότι το θέμα είναι λεπτό. Πολλοί λένε ότι σε όλες αυτές χώρες, αν αποκλείσουμε τη Μαλαισία και μιλώ για τη Μαλαισία για θρησκευτικούς λόγους, να είχα μία σχέση με τις αραβικές χώρες, αλλά να αποκλείσουμε τη Μαλαισία και τις αραβικές χώρες που έχουν ενεργειακούς πόρους, υπάρχει άποψη που ε, αναφέρει ότι το θρησκευτικό σκέλος πιέζει στα οικονομικά και την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά εάν θα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως αυτή τη λογική, ιδιαίτερα στον Ισλαμικό κόσμο, όπου γίνεται η άμεση προβολή του Κορανίου στο Σύνταγμα, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτή την πορεία. Και δεν θέλω να κρίνω τη θρησκεία. Απλώς θέλω να ε, ε, ρωτήσω κατά πόσο ο παράγων θρησκεία ε, έχει ειδικό βάρος στην αναπτυξιακή αυτή πορεία. Η κυρία Νέιτς. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας η οποία αποτελεί ε, τροφή για σκέψη για μας, για όλους τους συναδέλφους. Επειδή πιέζει ο χρόνος θα είμαι σύντομη. Από όσο γνωρίζω, πριν από 10 χρόνια το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών δημοσίευσε ένα πρόγραμμα για την αναπτυξιακή πορεία ιδιαίτερα του αραβικού κόσμου που συμμετείχαν και ακαδημαϊκοί διανοούμενοι και ούτω καθεξής. Και αν θυμάμαι καλά, ένα από τα βασικά ευρήματα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, είχε ως εξής. Ο αραβικός κόσμος είναι ελληματικός ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί δεν υπάρχουν δημοκρατικές δομές ενεργές ε, δημοκρατικές ε, δομές και οι γυναίκες αποκλείονται ως επιτοπλίστων από τη δημόσια ζωή. Υπήρχε και ένας τρίτος λόγος που τον οποίο δεν θυμάμαι. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που διέπει τις σχέσεις μας με τις διαφορετικές κοινωνίες του αραβικού κόσμου. Και όπως είπατε οι διάφορες ε, εκδηλώσεις του, της Αραβικής Άνοιξης προσέδωσαν μεγάλη ελπίδα σε αυτούς τους λαούς. Ίσως αναμέναμε πολλά και πολύ σύντομα. Αν ε, κάναμε μία αναδρομή στη δική μας ιστορία, στις επαναστάσεις στην Ευρώπη, κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, θα μπορούσαμε να δούμε πόσες επαναστάσεις απέτυχαν ικτρά καταρχήν και πόσο χρειάστηκε σε όλες τις περιπτώσεις, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να φτάσουμε σε μία σχετική σταθερότητα. Γι' αυτό η συσταλτική ερμηνεία της αρχής του More for More θα πρέπει να σχετίζεται με μία αναδρομή στο, στο παρελθόν. Έχουμε μία πολύ συσταλτική ερμηνεία και οπτική γωνία γιατί μιλάμε από ένα ολοκληρωτικό καθεστώς πρέπει να περάσει σε μια πλήρη δημοκρατία. Μα δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό σε ένα-δύο χρόνια, χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Γι' αυτό νομίζω ότι η προσέγγιση αυτή ε, ήταν ιδιαίτερα λανθασμένη. Ήταν κάπως πρωτόγονη. Εγώ συμμετείχα στην σύσταση της Task Force στην Αίγυπτο δύο χρόνια πριν και είδα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε ως προς την αρχή της αιρεσιμότητας ε, στην ε, Αιγυπτιακή κοινή γνώμη. Αν δείτε τον ε, τύπο της Αιγύπτου και τι ανέφερε, πώς αναφέρθηκε στην Task Force, δεν, γίνεται, δεν γινόταν πουθενά λόγος για την ρεσιμότητα. Είχε αποκριβεί. Και ένα από τα ε, αρεστά μου θέματα, θεωρώ ότι καμία δημοκρατία δεν μπορεί να ανθίσει χωρίς βιώσιμα πολιτικά κόμματα τα χρειαζόμαστε αν θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια μίας ε, λειτουργικής ε, δημοκρατίας. Και πολλοί διεθνείς οργανισμοί βοηθείας, ε, ιδιωτικοί ή δημόσιοι, δεν θέλουν να υποστηρίξουν ε, κόμματα τα οποία, δημοκρατικά κόμματα στα σπάργανα ακόμα, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι χρειάζεται πολύς χρόνος πριν φτάσουμε σε δημοκρατικά πολιτικά κόμματα. Θα ήθελα να σχολιάσετε. Ιδιαίτερα τη τελευταία μου σκέψη είναι σωστή και τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Σε Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά θέματα που ανακύπτουν από αυτή την άκρος ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα ήθελα να πω, με βάση αυτά που είπε η συνάδελφος για τη δημοκρατία, Νομίζω ότι είναι η ιδεολειψία μας, ε, η δική μας ιδεολειψία, το να θεωρούμε ότι η δημοκρατία θα επιτευχθεί την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη, την επόμενη εβδομάδα. Ιδιαίτερα εάν λάβουμε υπόψη ότι στον Ηνωμένο Βασίλειο οι γυναίκες μπόρεσαν να ψηφίσουν από το 1918 και μετά. Χρειάστηκε πολλούς αιώνες για να φτάσουμε σε δημοκρατικές δομές. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να σχολιάσετε ως προς τον αραβικό ε, σύνδεσμο. Τι είναι, ε, απλώς βγάζουν λόγους εκεί ή μπορεί πραγματικά να επιδράσει, γιατί δεν μου φαίνεται ότι μπορεί. Σε σχέση με τα κόμματα αυτά που βρίσκονται στα Σπάργανα, σε εμβριακή μορφή, επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι στην Αραβική Άνοιξη σε σχέση με άλλα μέρη του κόσμου, χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα με μεγάλη επιτυχία. Ίσως η ε, Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη καθώς και είπα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, αυτά τα μέσα ακριβώς για να επιδράσουν, για να δημιουργηθούν νέοι ηγέτες τύπου Ομπάμα. Ό,τι και να πείτε για την ε, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, έχει, Εκκλησία έχει έναν επικεφαλής ε, που ηγείται αυτή. Θεωρείτε ότι στο μουσουλμανικό κόσμο υπάρχει κάτι αντίστοιχο έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε ένα κοινό ρεύμα οι Σουνίτες και οι Σίτες, σε ένα κοινό σχήμα. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Δεν ξέρω κατά πώς υπάρχουν άλλοι που θα ήθελα να υποβάλουν ερωτήσεις. Α, η κυρία Γκόμες, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας θα ήθελα να σας ε, κάνω μερικά ερωτήματα. Ένα από τα προβλήματα στο παρελθόν Όταν επισκεπτόμεθα έργα που χρηματοδοτούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούσε η ε, υπηρεσία σας Εθνών στον Αραβικό κόσμο, βλέπε Ιράκ, Κάτι που μας στεναχωρούσε ήταν η χαμηλή ορατότητα ή προβολή της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράμματα του Οργανισμού Ανάπτυξης το ΟΗΕ. Μπορεί να υπήρχε κάποιος λόγος γι' αυτό, αλλά και κάποια πολιτική για να αποτραπεί η προβολή της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα έργα. Αυτό έχει αλλάξει και με ποιο τρόπο οι αραβικές εξεγέρσεις, η αραβική άνοιξη, είμαι βέβαιη ότι έκανε τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και τους οργανισμούς να προβληματιστούν, όπως κάναμε κι εμείς ε, στην πολιτική μας περισσότερο για περισσότερα και τα διάφορα μέσα που έχουμε. Αυτό πώς μεταφράζεται ε, σε χώρες όπου ο ανεξαρτήτως του επίπεδο διαβίωσης παραβιάζονται ή δεν γίνονται σεβαστά καθόλου τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα πιο θεμελιώδη από τους εκπροσώπους της εξουσίας. Um, I'm thinking about countries, for Οι χώρες του κόλπου, ε, ιδιαίτερα ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Τώρα φαίνεται να υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών στη Συρία. Οι περισσότεροι Άραβοι Σουνίτες δεν είναι, αν όχι όλοι. Υπάρχουν όμως και Σιητικές κοινότητες σε πολλές αραβικές χώρες. Αυτό πώς επηρεάζει τη δική σας δράση ως προς τη χρηστή διακυβέρνηση, την ανάπτυξη κτλ. Και ένα τελευταίο. Μόλις πριν από λίγο συζητούσαμε τη σύγκρουση μεταξύ μάλλον στην υπόθεση της Δυτικής Σαχάρας και γιατί δεν υπάρχουν καλύτερες σχέσεις και καλύτερη ένταξη. Και στο Μαρόκο και στην ε, Αλγερία. Τα ξέρουμε αυτά για το διεθνές δίκαιο και τα λοιπά, ότι είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών εσείς οι υπηρεσίες σας μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε με κάποιο τρόπο στη Δυτική Σαχάρα. Υπάρχει η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών η Μινούσο, αλλά η UNDP συμμετέχει με κάποιο τρόπο. Σε συμφωνίες, ας πούμε, τύπου Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου, εσείς έχετε ε, δυνατότητα να το ελέγχετε αν εφαρμόζονται ή όχι και αν είναι προ όφελο ή όχι του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Δόκτωρ Μπαούς, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι λένε τα σας τα σχόλια και τα ερωτήματα και θα προσπαθήσω να τα απαντήσω Το πρώτο ε, για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία και το ε, more for more, περισσότερα, με αντάλλαγμα περισσότερα. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τον αραβικό κόσμο, διότι άλλαξε και ο ίδιος ο αραβικός κόσμος. Δεν μπορούσαμε να συνεχίζουμε το παλιό πρόγραμμα. Όπως ε, αναφέρατε, θα τιμωρούσαμε άλλες χώρες που δεν ε, ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Ποιο είναι το κλειδί για όλα αυτά τα θέματα. Να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ελευθερία, στην κοινωνία των πολιτών και να βεβαιωθούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στις πολιτικές όλων των αραβικών κρατών και να υποστηρίζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και οι Ηνωμένε Πολιτείες αυτές τις προσπάθειες όλων της κοινωνίας των πολιτών, των κυβερνήσεων, των ε, ε, νέων ε, για να γίνεται όσο μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια και υποστήριξη. Εγώ τι έχω διαπιστώσει σήμερα. Στις περισσότερες αραβικές χώρες έχουν αλλάξει ηγεσίε, αλλά έχουν αλλάξει και νοοτροπία ηγεσίε. Διότι όλες οι ηγεσίε πλέον γνωρίζουν ότι ε, ο κόσμος στους δρόμους που έριξε την προηγούμενη κυβέρνηση, τον προηγούμενο πρόεδρο, θα τους ρίξει και αυτούς, αν δεν ανταποκριθούν στα αιτήματά τους. Άρα ακούν περισσότερο αφού όσο γίνεται με μεγαλύτερη ευαισθησία, τα αιτήματα και τις ανάγκες των λαών τους. Γι' αυτό θα πρότεινα κι εγώ ε, το Ένας από τους τρόπους εργασίας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ε, και με τους βουλευτές ε, περισσότερο και με τις ηγεσίες των χωρών και με οργανώσεις νέων πολύ περισσότερο διότι θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε όλοι ε, από πού έρχονται οι άνθρωποι αυτοί, τι ανάγκες έχουν και πώς το μεταλλασσόμενο περιβάλλον στην ίδια τους τη χώρα επιδρά στη ζωή τους. Για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή και την πολιτική δέσμευση. Το σημαντικότερο που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους είναι η παιδεία στον αραβικό κόσμο. Μέχρι τώρα η παιδεία πώς ήταν. Εντάξει, έχει βελτιωθεί το μορφωτικό επίπεδο, αλλά ποτέ η ποιότητα ε, της εκπαίδευσης και στα πανεπιστήμια και στα σχολεία στις αραβικές χώρες. Δεν υπάρχουν προγράμματα σπουδών, δεν διδάσκεται η δημοκρατία σε αυτά τα προγράμματα. Η κοινωνία από μόνη της είναι πατριαρχική, δεν έχει εκπαιδευτεί για θέματα δημοκρατίας. Ε, οι νέοι επίσης, μέχρι πολύ πρόσφατα, δεν ε, ήταν μια οντότητα ε, ε, αναγνωρισμένη, ξεχωριστή. Παρόλο που ο αραβικός κόσμος έχει τους περισσότερους νέους με τις περισσότερες ανάγκες, με τη μεγαλύτερη ενεργεία και τους περισσότερους νέους που θέλουν να μεταναστεύουν. Και σας το λέω από την ίδια μου την εμπειρία στα υψηλότερα επίπεδα που έχω εργαστεί και στον Αραβικό Σύνδεσμο και στον Αραβικό Κόσμο και στην Ιορδανία ότι η νεολαία χρειάστηκε να βρει στους δρόμους για να την προσέξουν, για να της δώσουν ε, σημασία. Συγγνώμη. Παρόλο ε, που πολλές εκθέσεις και του Αραβικού Συνδέσμου και των κυβερνήσεων έλεγαν ότι υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των νέων, ε, δυσφορία, χαμηλή ικανοποίηση, δεν εκπαιδεύονται σωστά, η παιδεία δεν συναντά τις ανάγκες της αγοράς και κάποια μέρα αυτό το σύνολο των νέων μπορεί να γίνει μια βόμβα ε, της νεολαίας και πράγμα που έγινε εν μέρη. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε και τους ενήλικες, αλλά έχει έρθει η ώρα να κοιτάμε και τα σχολεία, τους νέους μας, ε, τις πολιτικές για τους νέους και να βεβαιωθούμε ότι όλοι θα είναι ενταγμένοι. Και στα Ηνωμένα Έθνη, θα γνωρίζετε όλοι φαντάζομαι, ο Γενικός Γραμματέας ε, διόρισε ειδικό απεσταλμένο για την νεολαία, που είναι 28-29 ετών και προσπαθεί ε, να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να προωθεί σε αυτή την ιδέα ότι μπορούν και οι νέοι να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και να είναι τμήμα ε, της πολιτικής ζωής και ε, πραγματικά ο απεσταλμένος αυτός ταξιδεύει πάρα πολύ στην περιφέρεια του αραβικού κόσμου και είναι δύσκολη η δουλειά του γιατί τα θέματα που τον ενδιαφέρουν δεν απασχολούν τις κυβερνήσεις. Και αυτό θα πρέπει να το βοηθήσουμε. Επίσης, η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, άκρο σημαντική και αυτή. Η κοινωνία των πολιτών στον αραβικό κόσμο έχει κάποιες ρίζες, όχι πολύ γερές, όχι πολύ βαθιές και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ε, κλείσει αυτός ο κύκλος, αυτό το τρίγωνο κοινωνία πολιτών, κυβερνήσεις και λαοί. Ε, υπάρχει ζήτηση πλέον γι' αυτό, όχι κατά ανάγκη διότι δεν υπήρχε κοινωνία των πολιτών, αλλά γιατί τώρα έχουν αντιληφθεί το ρόλο της και πόσο αυτή μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες του κόσμου και να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Για τον Αραβικό Σύνδεσμο. Ήμουν αναπληρώτρια γενική γραμματέας ε, στον Αραβικό Σύνδεσμο μέχρι πριν από 18 μήνες. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι σημαντικό εργαλείο αυτή η οργάνωση, ένα σημαντικό θεσμός που μπορεί να βοηθήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις προσδοκίες ε, των αραβικών λαών να διεθνοποιήσει τα ζητήματα, να τα κάνει γνωστά. Μπορεί να υπάρχει κάποιο ζήτημα θεσμικών δυνατοτήτων ή κάποια άλλα θέματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να υποστηρίξουμε ε, τον Αραβικό Σύνδεσμο που με τη σειρά του προωθεί ε, τα μελήματα των πολιτών και τους μηχανισμούς έτσι ώστε να υπάρχει οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη μέχρι να υπάρξει κάτι διαφορετικό που δεν είναι του παρόντος, θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή τη σημαντική οργάνωση, αυτόν τον οργανισμό, την ανάπτυξη και η πολιτική ατζέντα είναι ρευστή και προχωράει. Σημειώνω αυτό που είπατε, ότι ορισμένοι θεωρούν ότι έχει χρεοκοπήσει, δεν νομίζω έχει ακόμα τη δυνατότητα επιρροή αν κοιτάξετε τις συγκρούσεις. Είχε λόγο ο αραβικό σύνδεσμος. Τώρα έχουμε και κοινό απεσταλμένο που προσπαθεί να λύσει τα ζητήματα στη Συρία. Πολιτικά εξακολουθεί να έχει ειδικό βάρος ο αραβικός σύνδεσμος. Δεν υπάρχει καμία διεθνής απόφαση που να λαμβάνεται ε, ερήμην του αραβικού συνδέσμου. Ακούνε και τους υπουργούς και τα ψηφίσματά του διαβάζουν και τον συμβουλεύονται. Είναι σημαντικό, θα πρέπει να στηρίζουμε τον Αραβικό Σύνδεσμο. Καθόλου δεν έχει ατονίσει. Είναι σημαντική η βοήθειά του και χρειαζόμαστε και εμείς ε, ως UNDP. Πιστεύουμε πολύ στην υποστήριξη των περιφερειακών οργανισμών. Έχουμε συμφωνία συνεργασίας με τον αραβικό κόσμο για να τους βοηθήσουμε ε, για την ε, οικοδόμηση δυνατοτήτων, παρακολούθηση εκλογών, ε, πύληση συγκρούσεων ε, και τα νέα προβλήματα του αραβικού κόσμου θα πρέπει να αντανακλώνται και στις εργασίες του αραβικού συνδέσμου, αλλά και σε αυτά που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΙΕ και όλοι οι εταίροι. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν κοιτάξουμε και πάλι την νεολαία, που σας είπα είναι η πιο πολυπληθής ομάδα του πληθυσμού, θα πρέπει να δούμε πώς ε, σκέφτονται, πώς δρούν, τι μέσα χρησιμοποιούν, ε, δρούν και κινούνται διαφορετικά από εμά. Αυτό είναι προφανές και θα πρέπει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο λειτουργούν οι νέοι και με τι ασχολούνται. Πρέπει να σας πω ότι η κόρη μου είναι 16 ετών και κάθε φορά που της λέω το παραμικρό μου λέει «Μα μαμά δεν με καταλαβαίνεις» δεν καταλαβαίνεις και τελικά το συνειδητοποίησα ότι δεν καταλαβαίνω τι θέλουν, πώς λειτουργούν, ούτε τι θέλει η κόρη μου, ούτε τι σκέφτεται, ούτε πώς σκέφτεται, ούτε τι ελπίδες έχει και προσδοκίες. Έχουν ε, άλλο κόσμο και άλλες ε, προτεραιότητες για την ανάπτυξή τους από εκείνες που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τους δώσουμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε και παγκοσμίω να ακούγεται η φωνή των νέων και να συμμετέχουν και στη χάραξη των πολιτικών και στα προγράμματα και στην εργασία και να χρησιμοποιούμε και τα δικά τους μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φτάνουμε σε αυτούς. Ελπίζω σύντομα να δούμε και βουλευτές στον αραβικό κόσμο που να είναι πολύ πιο νέοι στην ηλικία και να μπορούν πραγματικά να έρθουν στο προσκήνιο του πολιτικού γίγνεσθε και να υποστηρίζονται, να ψηφίζονται, να βγαίνουν εκλογές, ε, ε, βουλευτές, συγγνώμη, να εκλέγονται και βέβαια χρειάζεται μεγάλη επένδυση ε, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία, στην ειρήνευση να τα κατανοήσουν όλα αυτά οι νέοι και να τα ενστερνιστούν. Δεν ξέρω πώς να πω ε, το εξής και να σχολιάσω το θέμα των μουσουλμάνων και του Πάπα. Ε, στο μουσουλμανικό κόσμο δεν υπάρχει μία αρχή, ένας που να αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο του Πάπα. Ε, υπάρχουν θεσμοί όμως που ε, είναι σεβάσμοι, που, που θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, ε, να βοηθήσουμε να λυθούν τα προβλήματα. Το θέμα των Σούνιτων και των Σιητών στον αραβικό κόσμο. Εγώ στον αραβικό κόσμο μεγάλωσα. Ποτέ δεν ήξερα ποιος είναι Σουνίτης και ποιος είναι Σιήτης. Είναι μεγάλο το ζήτημα, αλλά είναι πολιτικό. Και έχει τόσο πολιτικοποιηθεί πλέον που θα πρέπει να προσέχουμε για το πώς το χειριζόμαστε όλοι. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι έχω την απάντηση και τη λύση, ούτε ότι έχω και το αντίδοτο, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στις πολιτικές και στα προγράμματα να βεβαιωνόμαστε ότι όλοι στον αραβικό κόσμο ε, θα πρέπει να σεβόμαστε τις μειονότητες και να ε, συμπεριλαμβάνονται όλοι στις διαβουλεύσεις. Έγιναν κάποιοι αποκλεισμοί στον αραβικό κόσμο σε κάποιους τομείς και τώρα πολιτικά πλέον ε, θα πρέπει να δούμε αυτά τα ζητήματα αλλά να βεβαιωθούμε ότι δεν θα εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση είναι πρωτοφανή αυτά τα φαινόμενα. Ποτέ δεν υπήρχαν στο παρελθόν στον αραβικό κόσμο μεταξύ των λαών, μεταξύ των πολιτών. Δεν είχα ακούσει ποτέ ότι οι Σίτες και οι Σουνίτες αλληλοσκοτώνονται. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό και θα πρέπει με τρόπο πάρα πολύ σοβαρό να το κοιτάξουμε πέρα και έξω από την πολιτική. Νομίζω ότι προσπάθησα να απαντήσω σε όσες ερωτήσεις μπορούσα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ για το χρόνο πρώτα απ' όλα που ε, αφιερώσατε και ήρθατε και ακούσατε ε, αυτά που είχα να σας πω, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε. Πραγματικά προσβλέπω σε μεγαλύτερη συνεργασία, ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, για να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε μια νέα πραγματικότητα στον αραβικό κόσμο και να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες για την ανάπτυξη, οι κοινωνικές, οι οικονομικές, ε, για να το κοιτάξουμε όμως από άλλο πρίσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μας. Ο διάλογος αυτός ήταν ωφέλιμος κατά διτό τρόπο. Μας προσφέρατε δύο θετικά, δύο πλεονεκτήματα με την παρουσία εδώ και την εμπειρία σας από το Ηνωμένα Έθνη ασφαλώς, αλλά και το γεγονός ότι εσείς που κατάγεστε από την περιοχή, γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα πράγματα που προσπαθείτε να μας μεταφέρετε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κανείς εμπλέκεται σε αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεται πόσο λίγο ξέρει την πραγματικότητα και πόσο ακόμα του μένουν να μάθει. Για τα παιδιά καλό είναι το ότι σκέφτονται. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που λειτουργεί το μυαλό τους και το ακονίζουν. Σας ευχαριστώ και εγώ. <clears throat> Και τώρα θέλουμε να απευθύνουμε στο τελευταίο θέμα μας. Είμαστε όλοι εδώ. Παρουσιάζουμε, όπως ξέρετε, την ενδιάμεση έκθεση για την παρακολούθηση της δίκης των δημοσιογράφων στην Τουρκία. Έχω μια ad hoc αντιπροσωπή εδώ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπα τον κύριο Βαλέντσα με πέντε δικούς μας συναδέλφους. Έχετε το λόγο κύριε Βαλέντσα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, η ομάδα αυτή ad ε, απαρτίζεται από μέλη της ε, Μικτής Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Τουρκίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση των δικών των δημοσιογράφων στην Τουρκία πάνω απ' όλα διότι υπήρξαν ε, κάποιες ανησυχίες και σαφείς ενδείξει ότι διώκονταν αυτοί οι δημοσιογράφοι για τα όσα είχαν πει και όσα είχαν γράψει και ενώ γνώριζαν οι δημοσιογράφοι, ενώ ο ισχυρίζονταν μάλλον η κυβέρνηση ότι ε, εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου ε, ήταν οι λόγια του οποίου είχαν ε, διωχθεί αυτοί οι δημοσιογράφοι, δεν μπορούσαμε να παραγνωρίσουμε τι υποψίε αυτέ. Γι' αυτό λοιπόν μετέβημε στην Τουρκία για να παρακολουθήσουμε αν γίνονταν κατά τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο αυτέ οι δίκε. Γιατί η ελευθερία του λόγου δεν θα πρέπει επουδεμνή να φημώνεται ε, για τους πολίτες ενός δημοκρατικού κράτους. Ως εκ τούτου ήταν ε, απόλυτα απαραίτητο για την ε, αντιπροσωπεία μας να γίνει αυτή η επίσκεψη. Πολλά πράγματα διαπιστώσαμε και αυτά επιβεβαιώνουν δυστυχώς τις ανησυχίες μας για την μερολεπτική δίκη, για το KCK αλλά και για το ODATV. Στις δίκες αυτές Κατηγορούνται οι δημοσιογράφοι διότι έγραψαν κατά τρόπο οργανωμένο ειδήσει ε, με στόχο την υποστήριξη ενός τρομοκρατικού σχεδίου ή σχεδίου τρομοκρατικής οργάνωσης. Αυτά όλα σε σχέση με άρθρα που έχουν δημοσιεύσει στον τύπο ε, βιβλία και φωτογραφίες που αξιοποιήθηκαν ως στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης συσχετισμού με τρομοκρατική οργάνωση και στις δύο περιπτώσεις η υπεράσπιστοι που υποστηρίζουν και οι ομάδες ε, για, την ελευθερία του τύπου. Ε, σημειώνω ότι πρόκειται για απλά σκηνοθετημένε δίκες και κατηγορίες στηριζόμενες μόνο σε εικασίες και χωρίς διαπίστωση συγκεκριμένων αδικημάτων ποινικών. Καταδικάζουν ως παράλογες αλλά και τραγικομικές τις κατηγορίες και τις δίκες. Ο ρόλος αντιπροσωπεία αντιπροσωπείας ad hoc βέβαια δεν ήταν να επιβεβαιώσει κάθε επιμέρους κατηγορία ή τα στοιχεία που τη στηρίζουν και τη συνοδεύουν. Σημειώνουμε ωστόσο τις επαναλαμβανόμενες ανησυχίες που εκφράζουν οι, δικηγόροι της, οι συνήγοροι της υπεράσπισης και οι ομάδες για την ε, υπεράσπιση των δικαιωμάτων ως προς την ε, αξιοπιστία των ε, στοιχείων που προβαλήθηκαν και στις δίκες KCK και στις δίκες ODA TV αλλά και άλλες δίκες τόσο χειρόγραφα άρθρων όσο και ε, βιβλία που έχουν και σε, μορφή ακόμη χειρογράφων τα βιβλία των δημοσιογράφων ήταν, είχαν κατασκευθεί από τις αστυνομικέ αρχές και είχαν αποτελέσει τη βάση του κατηγορητηρίου. Πολλές φορές το γεγονό ότι είχε πρόσβαση σε μια είδηση ο δημοσιογράφος πριν από τους συναδέλφους του και την είχε φυλάξει προκειμένου να αξιοποιήσει την ε, είδηση ε, χρησιμοποιήθηκε εις βάρος του. Ε, το KCK ε, θεωρήθηκε ότι με το να μην ε, δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικές με μία συγκέντρωση, η καταγγελία μιας προγραμματιζόμενης διαδήλωσης στην αστυνομία αποτελούσε σύμπραξη με το ΠΚΚ. Και έτσι ε, το άρθρο 12 του νόμου υπεριτύπου του 2004 αξιοποιήθηκε κατά τρόπον ακραίο. Υπήρξαν ε, επίσης ε, καταγγελίες που στηρίζονταν σε αρνητικές ειδήσει. Φερρυπίν τα προβλήματα που προέκυψαν μετά τον σεισμό στην πόλη Βάνα και η αρνητική, ο αρνητικός τύπος, τα, αρνητικά σχόλια που παρουσιάστηκαν χαρακτηρίστηκαν από τις αγγελικές αρχές ως αμάυρωση της εικόνας του τουρκικού κράτους. Ενώ οι αρχές ε, της υπεράσπισης με βάση την ε, ε, αλήθεια και τα συμφέροντα του κατηγορουμένου ε, έχουν παραγνωριστεί πλήρως. Η υποστήριξη λοιπόν στο μοντέλο του δημοκρατικού συνομοσπονδιακού κράτους ή τη περιφερειακή αυτονομία που επίσης υποστηρίζει το ΠΚΚ έχει χρησιμοποιηθεί ει βάρο των ε, αγωνιστών αυτών ή των, ε, των προσώπων που υποστήριζαν αυτέ τις ιδέες ως συνέργεια με τρομοκρατική οργάνωση. τηλεφωνικέ συνομιλίε και συνδιαλέξει έχουν ε, παρακολουθηθεί. Επίσης ε, σχέσεις μεταξύ δημοσιογράφων ή δημοσιογράφων και των απόρριτων πηγών τους αξιοποιήθηκαν από την εισαγγελία ενώ καταγγέλλονται από την υπεράσπιση ως παράλογες και κατασκευασμένες. Ε, Ένα από τους συνηγόρους υπεράσπισης στον, στη δίκη K KJK, Σημειώνω ότι θα ήταν ανθρωπίνω αδύνατο να διαβάσει τις χιλιάδες των σελίδων των απομακρυντοφωνημένων συνδιαλέξεων που αποτελούσαν τα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση του ODA TV, Υπάρχουν κάποιες λεγόμενες σημειώσεις από συνεδριάσεις οι οποίες ε, υποτίθεται πως έχουν τηρηθεί από τους κατηγορουμένους προκειμένου ε, να συγγράψουν τα βιβλία τους ή τα άρθρα τους και αξιοποιούνται εις βάρος τους. Ενώ ακόμη αμφισβητείται και η αυθεντικότητα τέτοιου είδους ε, αποδεικτικών στοιχείων. Στοιχεία σχετικά με ταξίδια στο εξωτερικό, φερειπίν θεωρήσεις διαβατηρίων, με τη σφραγίδα. Στη δίκη Κάτζεκα αποτελούν αποδεικτικά που υποστηρίζουν ε, το, τις κατηγορίες ότι κάποιοι από τους κατηγορουμένους είχαν μεταβεί στο Ιράκ για συνεμετοχή σε τρομοκρατικές ε, οργανώσεις. Ε, οποιαδήποτε δραστηριότητα δημοσιογράφων αποτελεί λόγο κατηγορίας. Μια άλλη ανησυχητική κατάσταση είναι η ύπαρξη των μυστικών μαρτύρων, των κρυφών ή ανωνύμων μαρτύρων, και βέβαια θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις δίκες των δημοσιογράφων στην Τουρκία για να διατυπώσουμε την τελική μας έκθεση το πρώτο εξάμεινο του 2014. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα της 18ης Απριλίου του 2013 για την, πρόοδο, για την έκθεση πρόοδου του για το 2012 της ε, Τουρκίας είχε σημειώσει ήδη ότι η αντιπροσωπεία ad hoc για την παρακολούθηση δικών δημοσιογράφων στην Τουρκία θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις δίκες ε, δημοσιογράφων και θα παρακολουθεί εκ του είναι και τη μεταρρύθμιση στο δικαστικό τομέα και την ελευθερία του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τις ανησυχίες του σε σχέση με τις εξελίξει δίκες και την πολύ μεγάλη περίοδο προσωρινής κράτησης πριν από την διεξαγωγή της δίκης που αφορά που και επηρεάζει πολλούς άλλους δημοσιογράφους και σκοπεύουμε βεβαίως να ασχοληθούμε και με τα θέματα αυτά. Ενημερωθήκαμε επίσης ότι ο ποινικό κώδικα της Τουρκίας και ιδιαίτερα ο αντιτρομοκρατικός νόμος αξιοποιούνται προκειμένου να διωχθούν ε, κάποιοι για δηλώσει που δεν έχουν καμία σχέση με τη βία, μόνο και μόνο επειδή υποστηρίζουν τους στόχους μιας ε, οργάνωσης ε, τρομοκρατικής. Επειδή τα άρθρα 26 και 28 του τουρκικού συντάγματος περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης ε, για λόγους δημόσιας τάξεως, εθνικής ενότητας και ασφάλειας κρατικής, πρέπει να παρακολουθήσουμε την κατάσταση προς τα άρθρα αυτά έτσι περαιτέρω. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι προηγούμενες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την κυβέρνηση της Τουρκίας για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου για την ελευθερία έκφρασης και την υποβολή της άνευ ε, χρονοτριβής στην ε, ευθεία γραμμή του ε, ε, της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Εθνών Δικαιωμάτων δεν έχει προχωρήσει. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσεως που έχει, που προωθήσει το ε, Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, το τελευταίο διάστημα και πάλι σε συμφωνία με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Εθνών Δικαιωμάτων που αποτελούν πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Σημειώνουμε ότι υπάρχουν πολλές δίκες εις βάρος και διώξεις βάρος δημοσιογράφος, ιδιαίτερα δημοσιογράφων εκείνων που ασχολούνται με το κουρδικό ζήτημα. Ήταν ε, επίσης δυσανάλογα υψηλή, υψηλά τα πρόστιμα τα διοικητικά πρόστιμα που επευλήθησαν σε, ορισμένα, ε, σε ορισμένες επιχειρήσεις ΜΜΕ που οδήγησαν έτσι στην ε, πολλές φορές ακόμη και στην πτώχευσή τους και το κλείσιμό τους, αλλά βέβαια και θέματα που έχουν να κάνουν με την ελευθερία στο διαδίκτυο. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε την κατάσταση, σημειώνουμε ότι η δέσμευση και η στράτευση του Υπουργού Δικαιοσύνης και τα ανώτατα ε, συμβούλια δικαστικών ε, λειτουργών της Τουρκίας ε, για συμμόρφωση με τις αρχές των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αποτελούν μια θετική εξέλιξη συνεχίζουμε το διάλογο που έχουμε αναπτύξει με τις τουρκικές αρχές και όπως είπα και νωρίτερα θα συνεχίσει η αντιπροσωπεία μας την παρακολούθηση των δικών. Μια προσεχής αποστολή προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα. Η τελική μας έκθεση θα κατευθεί στο πρώτο εξάμεινο του 2014. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Σοφοκλέους. Δεν πίστευα ότι θα με καλέσετε άμεσα, λέει ο κύριος Ντάρτμουθ. Θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος εξέθεσε πολύ σαφώς την κατάσταση για το τι συμβαίνει στην Τουρκία στην δίκη αυτών των δημοσιογράφων. Οι δίκες αυτές δεν ε, ανταποκρίνονται στα κριτήρια της δικαιοσύνης όπως την κατανοούμε εμείς. Και ε, λυπάμαι που δεν, που δεν είμαστε περισσότεροι για να ακούσουμε τι συμβαίνει. Γιατί οι συναδελφοί πιστεύουν στο μύθο ότι η Τουρκία και η κυβέρνηση Ερντογάν ε, συμμερίζεται τις ίδιες αξίες με τις δικές μας στην Υπηρετική Ευρώπη, διότι η Τουρκία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ και τέσσερα χρόνια, σε αυτή τη θητεία που βρίσκομαι εδώ, γίνεται λόγος για αξίες υπέρ της δημοκρατίας, κάτι που έφερε το Ηνωμένο Βασίλειο, διέδωσε στον κόσμο. Και θα ήθελα να πω προσωπικά και πατριωτικά ότι έτσι έχει κατάσταση. Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ τελειώνετε, λέει ο πρόεδρος. Και με αυτή την πατριωτική νότα θα ήθελα να πω ότι αυτές τις αξίες ε, τις συμμεριζόμαστε σε όλα τα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο, από το οποίο απέχει πόρο η Τουρκία. Θα ήθελα να καταστήσουμε σαφές στην Τουρκία ότι οι διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με βάση την συμπεριφορά της κυβέρνησης δεν έχουν καμία δυνατότητα επιτυχίας, καμία πρόπτικη, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Επίσης θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι τα προενταξιακά δάνεια προς την Τουρκία πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι ε, τα, τα φορτηγά της Ford δεν κατασκευάζονται πλέον ε, στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά στην Τουρκία με βάση ε, εύκολα δάνεια που χορηγούνται στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι πολύ φτωχή, απέραντη και διαφέρει πολύ ως προς αξίες που ακολουθεί και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα επιθυμούσα ο Πρωθυπουργό μου να μην μεταβαίνει την ε, Κωνσταντινούπολη και να λέει ακριβώς ότι ε, δεν πρέπει να υπάρχουν προσκόμματα στην προσχώρηση της ε, Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορώ να το δεχτώ. Τέλος, Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για αξίες τις οποίες δέχεται Εάν τις υποστηρίζει σοβαρά δεν μπορεί ούτε τώρα ούτε ποτέ να θεωρήσει, να λάβει υπόψη σοβαρά την προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαριστώ συνάδελφο για την εξαιρετική του εισήγηση. Όπως ξέρετε, Generosity στο έργο του, σε ένα σχετικό έργο και εφτά ήσαν ε, υπέροχοι, ε, προβάλλεται μια παρόμοια τάκα. Εν πάση περιπτώσει και εσείς μπορείτε να ε, υπερβείτε το χρόνο σας, αλλά από ένα λεπτό στα τρία η υπέρβαση είναι μεγάλη. Ο κύριος Σοφοκλέους έχει το λόγο. Καταρχάς, θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω με μια θέση θα έλεγα και με μια ευχή ότι η Τουρκία πρέπει να βρεθεί στον ευρωπαϊκό χώρο, να βρεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω ευχή γιατί δυστυχώς συμπεριφέρεται μέχρι αυτή τη στιγμή προσθέτοντας τα όσα έχουν λεχθεί και από την έκθεση η οποία παρουσιάστηκε θα τολμήσω να πω σκληρά ως εκβιαστής της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή από τη μια να θέλει να βρεθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια και από την άλλη να μην σέβεται ούτε τους θεσμούς, ούτε την ιστορία, ούτε την κουρτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την διεθνή νομιτάξη. Περιορίζομαι στο θέμα και να πω ότι είναι αδιανόητο μια χώρα η οποία θέλει να βρεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην σέβεται την ελευθερία του τύπου που αποτελεί κατάκτηση κάθε δημοκρατικής χώρας και προσθέτω στα όσα έχουν λεχθεί ότι η τελευταία Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων που εδρεύει στη Νέα Νιόρκη αναφέρει ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα παγκόσμια σε ρεκόρ αριθμό φυλακισμένων και έχω εδώ την έκθεση ότι είναι η πρώτη χώρα παγκόσμια που καταστέλει ουσιαστικά αυτό που κατακτήθηκε εδώ και πολλές δεκαετίες, την ελευθερία του τύπου. Είναι η πρώτη χώρα που ακολουθεί κακές πρακτικές για επιβολή της αυτολογοκρισίας σύμφωνα με τα όσα καταγράφει επαναλαμβάνω η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων. Και είναι η πρώτη χώρα που το 2012 έχει αυξήσει ουσιαστικά τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων. Δηλαδή μιλούν από μόνα τους τα στοιχεία. Αναφέρω τέλος ένα συγκεκριμένο παράδειγμα και κλείνω. Την περίπτωση της δημοσιογράφου Ροχάτ Εκμεξίν που για να είμαι πολύ πιο συγκεκριμένος που ξυλοκοπήθηκε άγρια γιατί δήθεν παρουσιαζόταν ως εγκληματίας, ληστής και ένοχος για ε, κλοπές που έχουν γίνει σε διάφορες περιοχές ενώ το πραγματικό της έκλημα είναι γιατί είχε μια ραδιοφωνική εκπομπή και εξέφραζε ελεύθερα τις απόψεις Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Νταφ, παρακαλώ. Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, μιλώ ως φίλος της Τουρκίας. Και πρέπει να σας πω ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι πρόσφατα ε, εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα στην Τουρκία και ε, έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ ε, η θέση του τύπου. Όχι μόνο οι δίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση από πλευράς του κυρίου Βαλένζα, από μας είπε τώρα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει επεκταθεί αυτή η ιστορία και πέρα από τις δίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το κοινοβούλιο μας θα πρέπει να τα παρακολουθεί πολύ στενά αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Ερντοάν και το κυβερνών κόμμα πιέζουν κατά τέτοιο τρόπο τους δημοσιογράφους και τους ε, ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, ώστε αυτοί ε, εμφανίζουν ένα ιδιαίτερο αυξανόμενο φαινόμενο Αυτολογοκρισίας. Και μάλιστα γίνονται όργανα και φερέφωνα πλέον αποκλειστικά ε, της ιδεολογίας ε, του ΑΚΠ. Πού είναι η πολυφωνία που είχαμε κάποτε στην Τουρκία. Και μάλιστα ε, με έναν τύπο πάρα πολύ επικριτικό πολλές φορές και οξύνου. Βλέπετε τι έγινε στην υπόθεση Γουλέν και τη σύγκρουση με ε, το ΑΚΠ και ε, τι αντίκτυπο έχει αυτό στην εφημερίδα Ζαμάν και στην Τουρκία. Στοχοποιείται από την κυβέρνηση. Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμα ατυχές που συμβαίνει. Στο εξής. Ο Πρωθυπουργός Ερδοάν φαίνεται ε, ότι κατασκευάζει δημοσιεύματα στον τύπο που είναι τελείως παράλογα ορισμένα, όπως η κατηγορία ότι το Ισραήλ κρυβόταν πίσω από το πραξικόπημα στο Κάιρο. Και μετά αρχίζει να πιστεύει τα ίδια τα δημοσιεύματα που κατασκεύασε ο ίδιος. Και αυτό είναι αρκετά σοβαρό και αρκετά επικίνδυνο. Όσο και ασυνάρτητο, δεν συνάδει με το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φλότρο που είναι μία από τα μέλη της αντιπροσωπείας. Μικρόφωνο κυρία Φλότρο. Να μένω, κανονικά δουλεύει, εν πάση περιπτώσει. Ακούγομαι τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα νέο εργαλείο, ad hoc αντιπροσωπεία. Για ποιο λόγο? Όχι για να κατηγορήσουμε και μονομερός να στραφούμε κατά των τουρκικών αρχών, όπως ακούω από συγκεκριμένου συναδέλφους. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτή η πρόθεσή μου. Το λέω. Γιατί και ο πρόεδρος Βαλέσα... Δεν δουλεύει αυτό το μικρόφωνο, μάλλον πρέπει να αλλάξει ο μιλήτρια. Παρακαλώ, ε, αλλάξτε μικρόφωνο γιατί δεν δουλεύει αυτό. Λοιπόν, έλεγα σύντομα ότι έχουμε ένα νέο μέσο τώρα, ad hoc αντιπροσωπεία μετά από τροπολογία της δικής μου ομάδας το, τότε, πριν από 1,5 χρόνο, όταν ε, ανησυχούσαμε βαθύτατα σε σχέση με την ελευθεροτυπία στην Τουρκία και την ελευθερία της έκφρασης γενικότερα. Η αποστολή αυτής της αντιπροσωπείας δεν ήταν, όπως άκουσα από ορισμένους συναδέλφους, να ε, κατηγορήσει τις τουρκικές αρχές ε, μονομερός και μεροληπτικά. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, ούτε η δουλειά του συναδέλφου Βαλένσα που ήταν επικεφαλής. Αλλά αυτό που θέλαμε ήταν να δείξουμε το στένος μας ότι προσοχή, σας παρακολουθούμε μονίμως, όχι μόνο όταν ερχόμαστε με τις αντιπροσωπείες και με τις εκθέσεις, παρακολουθούμε πάγια αυτό το θέμα που είναι και ο ακρογωνίος λήθος της δημοκρατίας, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθεροτυπία με ποια προοπτική, την προοπτική βεβαίως να διατυπώσουμε τις καλύτερες δυνατές συστάσεις και να ασκήσουμε απέναντι στις τουρκικές αρχές αλλά και το σύνολο των παραγόντων που συμμετέχουν ε, στην πολυφωνία και τον επαγγελματισμό του τύπου στην Τουρκία ε, τις συστάσεις μας. Ωραία. Πρέπει να πω τώρα ότι από αυτή τη σκοπιά τα σχόλια που ακούσαμε από κάποιους συναδέλφους ε, μπορούν να μας κάνουν να λυπηθούμε για αυτή την πρωτοβουλία. Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα, νομίζω, ως βουλευτές να δούμε εμείς τι μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους αυτούς, γιατί είναι πολλοί, εξακολουθούν, είναι πάρα πολλοί όλοι αυτοί. Το ξέρουμε, τους βλέπουμε μέρα με τη μέρα, οι οποίοι στην Τουρκία διαδηλώνουν υπέρ της δημοκρατίας, των ελευθεριών και την ελευθερία του τύπου η έκθεση επισημαίνει κάποια κατάφορα ζητήματα, ακόμα και αν είναι έκθεση του 2012. Έκτοτε έχουν συμβεί πράγματα και θα πρέπει και πάλι να μετρήσουμε τον αντίκτυπο. Ε, βλέπετε το τέταρτο πακέτο ε, των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη. Επίσης υπάρχει και αυτό το θέμα το κουρδικό ζήτημα. Γιατί το κουρδικό ζήτημα και πώς αντιμετωπίζεται το θέμα της ασφάλειας ε, και το κουρδικό μέσο των αντιτύπων των τρομοκρατικών νόμων είναι καθοριστικό ζήτημα και για τον τύπο και για τους δημοσιογράφους στην Τουρκία. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συγκεντρώνει την προσπάθειά μας, την προσοχή μας και τη βοήθειά μας. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να υποστηρίξουμε αυτή την ειρηνευτική προσπάθεια, αγαπητοί βουλευτές. Και κάτι άλλο, αλλά αυτό θα το κάνουμε στις επόμενες αντιπροσωπείες, είναι η ε, υπόθεση του πάρκου Γκεζή και, και αντίκτυπο που έχει. Γιατί άνοιξε τα μάτια ε, των πολιτών, ως, των Τούρκων, ως προς την ε, κατάσταση του τύπου στην Τουρκία. Πολύ γρήγορα, γιατί σε διάφορα ραδιόφωνα κανάλια, σε γη εφημεριδες εφημερίδες, 5-6 μέρες διαδηλώσεις, σιωπή. Ενώ σε άλλες ε, τηλεοράσεις 24 ώρες το 24ωρο non-stop εικόνες που βλέπουμε συνεχώς. Προβοκάτορες της αστυνομίας που πηγαίνουν ε, με τους ταραξίες και διάφορες χειραγωγήσεις. Τα ξέρουμε αυτά. Δηλαδή, με ποιο τρόπο χειρίζονται ή διαχειρίζονται την πληροφορία, ε, η αυτονόμηση και η ανεξαρτησία. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα από πίσω ή το ΑΚΠ ή κάποιο λόμπι στα μέσα ενημέρωσης. Το ζήτημα που μας ενδιαφέρει είναι να αυτονομηθεί ε, η δημοσιογραφία, ο τύπος και οι δημοσιογράφοι. Μια αυτονομία, μια αυτοτέλεια με επαγγελματισμό, με διάρθρωση. Ε, να υπάρχει πραγματικά επάγγελμα δημοσιογράφος στη Δουρκία και να βλέπουμε και ποια είναι η χρηματοδότηση του τύπου ε, είναι ε, ο πρόεδρος διακόπτη. Τελειώνω, τελειώνω. Είναι πολύ πολλωμένη λοιπόν η κατάσταση και μια προσωπικότητα αρκετά αυταρχική όπως είναι αυτή του Πρωθυπουργού που έκανε ε, αυτά τα δημοσιεύματα για την ε, προπαγάνδα και ε, αυτά τα συνωμοσιολογικά που είπε και ο Άντρου Ντάφ και τα κυκλοφόρησε στον τύπο, δεν έχει καταλάβει και ο κόσμος. Αλλά το θέμα είναι να αυτονομηθούν οι δημοσιογράφοι, να χειραφετηθούν στην Τουρκία. Και αυτή θα πρέπει να είναι η βασική μας ανησυχία και το μέλημά μας ε, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Uh, Νομίζω ότι ε, ε, έχετε δίκιο, ότι ακούσαμε μάλλον αυτό που θέλετε να πείτε, η κυρία Γκόμες. Καταλαβαίνω τις ε, ανησυχίες σας ε, για τη... και τους φόβους που έχουν εκφραστεί σε σχέση με την ε, προσχώρηση, ενδεχόμενη προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω όμως ότι η αποστολή, η μας πρέπει να συνεχιστεί. Επειδή συναντήθηκα με πολλούς θαραλέους ανθρώπους στην Τουρκία που τάσσονται υπέρ της ελευθεροτυπίας, της ελευθερίας του λόγου, υπερασπίστηκαν το πάρκο Γκεζή. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν αυτό τον αγώνα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν. Η Τουρκία πάντα θα είναι εκεί, είναι ο γείτονάς μας, είναι ο εταίρος μας και πρέπει να υπερασπιζόμαστε εκείνους που υποστηρίζουν το δικαίωμα λόγου. Τα η Τουρκία που είναι μια μεγάλη χώρα κινείται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση όπως δείχνει η ενδιάμεση έκθεση και τώρα μας απασχολεί η αυτονομία της δικαιοσύνης. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πια μια κοσμική Τουρκία υπό την κυβέρνηση Ερντογάν. Εγώ είχα επικρίνει την έλλειψη ελευθεροτυπίας και το δικαίωμα επίκρισης της ε, στρατιωτικής ε, επικυριαρχίας ε, και κατοχή στην Κύπρο, καθώς και άλλων και μαλικών στοιχείων μέσα στα πλαίσια του βαθέως κράτους. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι το ΑΚΠ βρίσκεται μακριά από τους κεμαλιστές, αλλά δεν υπερασπίζει την, την ε, δημοκρατία, με συγχωρείτε. Επίσης υπάρχει υποστήριξη της Συρίας και του Ιράκ ε, συγκεκριμένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Και όπως είπε ο Άντριου Νταφ από τους φιλελευθέρους, η ιδέα του Ερντογάν ώστε στρατιωτική στρατηγή ε, να λαμβάνουν και λαμβάνουν εντολές από το Ισραήλ είναι κάτι το γελίο. Επίσης το γεγονός ότι δεν θα ε, ανοίξει η ερατική σχολή της ε, για τους χριστιανούς και τους Ορθοδόξους μας δείχνει ότι δεν υπάρχει πια καμία εγγύηση στην Τουρκία. Ε, κύριε ε, Βαλέσαν, αν θέλετε να συνοψίσετε με μία πρόταση. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, θα τα λάβω υπόψη, αλλά θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πολλά θα πρέπει να γίνουν από πλευράς Τουρκίας. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι οι τουρκικές αρχές θέλησαν να συνεργαστούν μαζί μου και με την αντιπροσωπεία. Θα ήθελα κάπως να ε, να απαλύνω τις εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί και η διάσκεψη, στη διάσκεψη των Προέδρων είπαμε ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για την ελευθεροτυπία, για τους φυλακισμένους δημοσιογράφους και ούτω καθεξής. Εκεί θα αρκεστούμε, δεν θα μιλήσουμε για την μελλοντική προσχώρηση, ενδεχόμενη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχω μια συγκεκριμένη αποστολή την οποία και θα ακολουθήσω. Ευχαριστούμε πολύ και με... Και έτσι ολοκληρώνουμε τη συνεδρία σήμερα. Θα τα πούμε στις 23-24 Σεπτεμβρίου την προσεχή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας.